Chers collègues, notre rapport... Αγαπητοί συνάδελφοι, η εισηγητριά μας είναι παρούσα. Άρα μπορούμε να αρχίσουμε τις εργασίες μας, αν θέλετε. Et ainsi nous... Και μπορούμε να εξτάσουμε το σημείο 8 της μελίστας διάταξης, όπου η αντιπρόεδρο τον Άντια θα μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησή για τις 20 κύριες ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων σχετικά με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Παρακαλώ, η συγκήτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σαν Επιτροπή Απασχόλησης είχαμε Ε, να εξετάσουμε αυτά στις 20 κύριες ενισχύες για την ε, ενιαία αγορά, θέματα υγείας κλπ. που ε, μπήκουν στις δικές μας αρμοδιότητες. Θα φαντάσετε βέβαια ότι είναι πολύ δύσκολο να συνενώσει καταρχήν κάποιο από τις, τις ανησυχίες αυτές σε μία σελίδα και γι' αυτό χαίρομαι ότι μπορούμε με τις τροπολογίες να δώσουμε περισσότερη ζωή σε αυτό το θέμα γιατί εγώ τις έχω απλώς και αγραφήσει έκανα την κατανομή αυτή σύμφωνα με τα θέματα. Θα μπορείτε να δείτε το θέμα της ε, κοινωνικής ασφάλισης και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που με ανάγκασα να εξετάσω το θέμα της κοινωνικής προστασίας περισσότερο προσεκτικά, γιατί ξέρετε αγαπητοί συνάδελφοι και εσείς έχετε ακούσει φυσικά από πολίτες ε, επερωτήσεις, επιστολές κλπ. ότι το σύστημα δεν λειτουργεί, ιδίως αν κάποιος μεταβεί σε μια άλλη ε, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εργαστεί εκεί. Και επίσης δεν υπάρχει ο σωστός συσχετισμός με την ε, ασφάλεια ανεργίας, επιδόματα ανεργίας. Είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή αυτές οι διοικητικές διαδικασίες είναι πολύ διαφορετικές από χώρα σε χώρα και θα πρέπει κανένας να έχει πρόσβαση σε διαφορετικές ε, υπηρεσίες και δεν απορώ λοιπόν που πολλοί πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, διστάζουν να εκμεταλλευτούν την ελεύθερη κυκλοφορία. Θέλουμε λοιπόν να πούμε ότι θα πρέπει να ξαναξεκινήσει η συζήτηση που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια και να σκεφτούμε ότι αν κάποιος ξέρει πραγματικά ότι τα επόμενα ας πούμε 10 χρόνια, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, θα κινείται μεταξύ διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια θα εργάζεται στο ένα κράτος, μια στο άλλο, μήπως υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει ένα ξεχωριστό σύστημα κοινωνικής προστασίας. Δεν ξέρω ποια μορφή θα μπορεί να έχει κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχουν πολλές δυνατότητες, αλλά όποια μορφή και αν έχει είναι κάτι που αξίζει οπωσδήποτε να συζητήσουμε και μάλιστα να γίνει μια πολιτική συζήτηση πάνω σε αυτό, γιατί η ακαδημική συζήτηση έχει ήδη γίνει και διαφοροποιημένα. Αλλά ακριβώς αυτή τη στιγμή που προσπαθούμε να προωθήσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία, που βλέπουμε την αναγκαιότητα για την καταπολέμηση της ανεργίας, να υπάρχει δυνατότητα εργασία σε μια άλλη χώρα μέλος, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της εξασφάλισης της εκμετάλλευσης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προωθήσουμε εκείνοι που εργάζονται ίσως μια μόνο φορά σε ένα άλλο κράτος μέλος να έχουν πιο απλές διαδικασίες, να είναι πολύ πιο εύκολο να συνυπολογιστεί ο χρόνος εργασίας κλπ. Τελευταία τελικά έχουμε μία πρόταση για μία προσέγγιση μοναδικής ε, θηρίδας γιατί όταν μεταβεί κάποιος σε μια άλλη χώρα δεν χρειάζεται μόνο την θέση απασχόλησης του θα πρέπει να δει πώς θα ασφαλιστεί όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πώς θα μπορέσει να δηλωθεί στην κοινότητα, να αλλάξει το αυτοκίνητο της πινακίδες κλπ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πολίτης είναι ο πελάτης και αυτός ο πελάτης, ο πολίτης δηλαδή, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μιας μονοθερητικής πρόσβασης για να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Στο σημείο 4 και 5 αφορούν ε, όλα τα θέματα της ε, ασφάλισης υγείας, της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Υγείας που ξέρετε ότι χρειάζεται ακόμα περισσότερη ενημέρωση. Θα πρέπει και εκεί να κληθούν τα κράτη-μέλη να διαθέσουν τις σχετικές πληροφορίες και κυρίως η επιστροφή του κόστους περίθαλψης να γίνεται γρήγορα και απλούστερα. Οι τομείς 6 και 7 αναφέρουν τις ε, επαγγελματικές ε, ε, γνώσεις και τις, την μετεκπαίδευση ή εκπαίδευση γενικά και τονίζουμε μια θέση που είχαμε πάρει και στο παρελθόν και θέλουμε να προτείνουμε να είναι πιο γλίγορη, πιο απλή η αναγνώριση, αλλά όχι μόνο η τυπική αναγνώριση, αλλά και η ανεπίσημη. Ένα σημαντικό σημείο είναι η μηδενική ανοχή για ε, διακρίσεις που θα πρέπει να ισχύσει όλα τα κράτη-μέλη. Και αναφέρεται το θέμα των εργαζομένων και την απόσπαση των εργαζομένων, που είναι ένα θέμα που εξετάζεται έντονα τις τελευταίες εβδομάδες, είναι το θέμα της σύνταξης. Δηλαδή όταν πάω εγώ σε μια άλλη χώρα μέλος, θα πρέπει να έχω την εγγύηση ότι στο τέλος ε, της ε, ζωής, της ζωής, ε, να μην ε, υποφέρω επειδή έχω εργαστεί σε διάφορες χώρες μέλη. Δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο και εδώ θα πρέπει να υπάρχει ε, η σωστή δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιδοτικών δικαιωμάτων. Αυτές είναι οι σύντομες ε, παρατηρήσεις, λίγα σημεία. Υπάρχουν πολλά θέματα βέβαια που παίζουν ρόλο και θα χαρώ να υπάρχει έντονη συζήτηση με πολλές τροπολογίες για να δώσω περισσότερη ζωή γιατί έχουμε βέβαια το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, υπάρχει αυτό, αλλά η πραγματικότητα διαφέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Η συγκίτρια μας υπενθύμησε τους περιορισμούς κατά τους οποίους δρούμε. Είμαστε ανεπίσημα εδώ συνδεδεμένοι είσαστε αναγκασμένοι να έχετε ένα σύντομο κείμενο και η πρόταση που κάνετε καλύπτει τις ε, πέντε ε, προτάσεις πάνω στις οποίες θα μπορούσε να αναπτυχθεί η δική μας ε, Επιτροπή και να υποβάλει σχετικές προτάσεις στον κύριο συγητή που είναι στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Λοιπόν, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον σκιώδη συγητή της Κομισιόν καταρχήν και μετά ως συγγήτρια στη μια μεγάλη επιτροπή για το θέμα αυτό. Η κυρία Λοπέα Φωτανιά και μετά η κυρία Στάνμπρουκ. Ευχαριστώ. Όντως, Πρόεδρε, νομίζω ότι κατέβαλε ήδη την προσπάθεια συγγήτρια για να κατανοήσει και να συλλέξει την ουσία των ζητημάτων που μας ενδιαφέρουν και που παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην εσωτερική αγορά. Φυσικά αν θέλουμε να κάνουμε μία πραγματική ένωση και οι εργαζόμενοι να δίνονται να εργαστούν σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά χρειάζεται να βελτιώσουμε σημαντικά την κατάσταση στην Ισπανία. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλούς νέους που επιθυμούν να εργαστούν και μεταβαίνουν σε άλλες χώρες και συνεχώς υπάρχουν παράπονα ε, ότι σε κάποιες χώρες να δουν περισσότερα προβλήματα από ό,τι σε άλλες ε, το λέω αυτό διότι θα πρέπει να υπάρξει μια, ε, μια βελτίωση της όλης κατάστασης. Λοιπόν, στο σημείο 1 θα πρέπει να συζητήσουμε σημαντικά σχετικά με το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο και όπως αναφέρω θα πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά. Επίσης, ε, τουλάχιστον στην ισπανική εκδοχή, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταστήσουμε σαφέστερο αυτό το οποίο ζητάμε. Στο σημείο 7 μιλάμε για το θέμα των ε, συγκρίσιμων προσόντων ε, και είναι πολύ σημαντικό το θέμα στην, Ιταλία, στην Ισπανία αυτή τη στιγμή. Οι εργαζόμενοι μπορεί να μεταβούν σε μια χώρα όπως ε, στην Ισπανία όπου κάτι που πολύ συχνά συμβαίνει χωρίς πολλά εμπόδια αλλά δυστυχώς σε άλλα κράτη αντιμετωπίζουν πολλούς φραγμούς, πολλά εμπόδια διότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτής της συγκρισιμότητας και της αναγνώρισης ε, των σπουδών. Τώρα, σε ό,τι φορά τις ε, διακρίσεις, ε, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα, θα πρέπει να διευκρινίσουμε τι ακριβώς ζητάμε για τις πολιτικές που συχνά μπορούν ε, να οδηγήσουν σε διακρίσεις. Πάντως ε, κρίνω ότι η έκθεση είναι σωστή. Φυσικά σε μια σελίδα δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλα όσα επιθυμούμε. Πάντως ε, με ορισμένες τροπολογίες αναμφίβολα μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω ένα ήδη καλό κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Στάινρου και μετά κυρία Μπαστός. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγητρία για την γνωμοδότηση. Το έγγραφο εργασίας της που ήταν η βάση αυτής της γνωμοδότησης δεν είναι ικανοποιητικό. όσον αφορά τις ανησυχίες των πολιτών και των επιχειρήσεων για την ιστορική αγορά, γιατί δεν προτείνει λύσεις και επαφείται άρα σε εμά ε, να το κάνουμε. Και ως εισηγήτρια των ε, σοσιαλδημοκρατών σύμφωνα σε μεγάλο βαθμό με αυτά τα οποία ανέφερε η εισηγήτρια και η κυρία Λόπες αλλά πρέπει να ενισχυθεί το κομμάτι βεβαίως των εργαζομένων και των εργασιακών ε, δικαιωμάτων. Καλό το ότι αναφέρατε την οδηγία περί απόσπασης και αν δούμε τις βασικές 20 ανησυχίες για την εσωτερική αγορά και εμείς η Επιτροπή μας πρέπει να πει πως ε, πρέπει κάτι να κάνουμε για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων εργαζομένων και εδώ πέρα δεν είναι βεβαίω όλες οι κύριες ανησυχίες ε, υπάρχουν παραδείγματος χάρη οι δημόσιες προμήθειες ε, διοικητικά εμπόδια, χωρίς βεβαίως να παραμελήσουμε και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γι' αυτό καταθέσαμε, θα καταθέσουμε κάποιες ε, τροπολογίες ε, για να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση της εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, το θέμα των δημοσίων συμβάσεων ε, είναι ένα από τα 20 συζητήματα ε, αν πάρουν δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της δικής μας Επιτροπής, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί το ζήτημα της κατανομής των αρμοδιοτήτων που, καθορίσαμε, που ορίσαμε με την Επιτροπή ΙΜΚΟ, αλλά εν πάση μπορούμε ούτως ή άλλως ε, να εκφραστούμε επί του ζητήματος, διότι το θέμα των κρατικών προμηθειών ε, μπορεί να ακολουθήσει μια συζήτηση που ήδη είχαμε, όταν η τελευταία έκθεση αναφορικά με τις κρατικές προμήθειες ε, συζητήθηκε. Μια έκθεση νομίζω πως δεν θυμάμαι ποιος ήταν η συγκεκριά. Είχαμε τη συζήτηση σχετικά με τη συζήτηση κοινωνικής ρήτρας ε, στο ζήτημα των δημοσιοβιβάσεων. Κυρία Μπαστός που είναι η συγκήτρια επί στην Επιτροπή ΙΜΚΟ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγητριά μας ε, για την γνωμοδότηση. Αναφέρθηκαν και οι προαλήσαντες συνάδελφοι, ειδικά τις διάφορες φάσεις ε, που πέρασε η γνωμοδότηση η οποία κατόρθωσε να συνοψίσει τα σημαντικά ζητήματα τα οποία απασχολούν την Επιτροπή μας ε, επί των σημαντικών αυτών ζητημάτων που απασχολούν και προβληματίζουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα ήθελα να πω πως ως επί της ουσίας ε, στην Επιτροπή ΙΜΚΟ η στρατηγική είναι μια στρατηγική η οποία δεν θέλει να βρει ε, συγκεκριμένη λύση για κάθε μία, καθένα από το προβληματισμό των ε, πολιτών. Όχι, θέλουμε να δώσουμε κατευθυντές γραμμές και προσανατολισμούς, ειδικά προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να υποδείξει τα κατάλληλα νομοθετικά βήματα τα οποία πρέπει να αναλάβουν τα κράτη-μέλη. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν η πολιτική βούληση ε, ώστε να επιληθούν ζητήματα που συχνά είναι θεμελιώδη και που απασχολούν ε, καθημερινά τους πολίτες και αυτό τους οδηγεί να έχουν ε, μια δυσπιστία απέναντι στην ενιαγωρά. Πάντως, ε, μετά από τις αναλύσεις που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά αυτά τα οποία συζητήθηκαν και στην αρμόδια Επιτροπή, υπάρχουν τρεις βασικές ελλείψεις ε, που οδηγούν ε, σε αυτές τις ανησυχίες, τον προβληματισμό των πολιτών αναφορικά με τη λειτουργία της ιστορικής αγοράς. Το πρώτη αφορά την ενημέρωση. Οι πολίτες δεν γνωρίζουν τα, δικαιώματά τους. Δεν γνωρίζουν που πρέπει να αποτανθούν ε, και πολλές φορές ε, δεν κατανοούν επαρκώς ε, τα πλεονεκτήματα από τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Και δεν έχουν και τα σχετικά ωφέλη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, κάποιες εκστρατείε ε, ευαισθητοποίησης, πληροφόρηση. Αυτή η γνωμοδότηση της συναδέλφου Χίρσου ε, καταδεικνύει αυτήν την, ε, αυτόν τον προβληματισμό των πολιτών. Υπάρχουν ζητήματα πολύ απλά, όπως τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης, της κοινωνικής πρόνοιας για τους προλήτες που πρέπει, να εργαστούν σε ένα άλλο κράτος μέλος να γνωρίζει ποιες είναι οι διαδικασίε διαδικασίες που αφορούν την κατοικία, διαμονή κλπ. Επίσης το θέμα του συντονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης ε, με συγκρίσιμα προσόντα. Ε, κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά την καθυστερημένη ε, μεταφορά στα εθνικά δίκαια των οδηγιών. Συνεχίζουν να υπάρχουν μια σειρά από διαδικασίες, από προσφυγές κατά κρατών μελών για την καθυστερημένη μεταφορά οδηγιών στον εθνικό, εθνική νομοθεσία. Αυτό λοιπόν οδηγεί όπως καταλαβαίνετε σε δυσκολίες ε, τις οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες μας. Ε, οι πολίτες λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν ε, πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά την κινητικότητα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μέχρι τώρα. Πολλές φορές αναγκάζονται να παραιτηθούν από κάποιες ε, δραστηριότητές τους, διότι έχουν άγνοια και η τελευταία έλλειψη είναι νομοθετικής φύσης. Συχνά Υπάρχουν προσδοκίες από πλευράς ε, των πολιτών ε, και των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων, που πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πάει παραπέρα σε ό,τι αφορά τα νομοθετικές εξουσίες. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Και αυτό που με απασχολεί είναι να υπάρξουν πολιτικοί προσανατολισμοί και να υπογραμμίσουμε την ε, πολιτική βούληση των κοινωτικών οργάνων αλλά και των κρατών μελών έτσι ώστε να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, να ξεπεραστούν αυτές οι ελλείψεις και να δώσουμε τις απαραίτητες απαντήσεις τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε μια κρίση. Η ιστορική αγορά προσφέρει δυνατότητες για την υπέρβαση αυτής της κρίσης. Τώρα επανερχόμενη στο θέμα της ε, γνωμοδότησης ε, της Επιτροπής Απασχόλησης ε, που θα συμπεριληφθεί και στην τελική έκθεση της, της Επιτουσίας Αρμόδιας επιτροπής θα πρέπει να τονίσουμε το ζήτημα της ε, μονοευθυντικής στηρίδας, ώστε ο πολίτης ε, με τρόπο απλό και γρήγορο να επιλύει όλα τα διοικητικά προβλήματα και ζητήματα. Επίσης το ζήτημα της δυνατότητας μεταφοράς της κοινωνικής ασφάλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για να υπάρχει μια πιο απλή πρόσβαση στην αγορά εργασία. παράλληλα φυσικά με την αναγνώριση των προσόντων. Πολλά ακόμα θα μπορούσα να προσθέσω, αλλά προ το παρόν αρκούμε σε αυτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια. Ναι, κυρία εισηγήτρια, σωστά, δεν το είπα. Επί τη ουσία, εισηγήτρια. Προτού να δώσω το λόγο στην δική μα εισηγήτρια, θα ήθελα να συμπληρώσω αυτό που είπε η κυρία Στάινρουκ και να αναρωτηθώ σχετικά με την φύση αυτού του εγχειρήματο. Ε, υπήρξε η λευκή βίβλος του κυρίου Μόντι, υπήρξε ε, η βίβλος, δεν ξέρω θυμάμαι ποια τη χρώμα είχε, του κυρίου Μπαρνιέ. Τώρα υπάρχει, ε, υπάρχουν αυτές οι 20 προτάσεις και αυτές οι 20 προτάσεις καθορίζονται από μια προσέγγιση αναφορικά με τα διακυβεύματα της ιστορικής αγοράς όταν διασχίζουμε τα σύνορα. Όταν μιλάμε για την εσωτερική αγορά στους πολίτες μας, ε, το ζήτημα το οποίο τίθεται δεν είναι τι συμβαίνει όταν διασχίσουν τα σύνορα, διότι κάθε μέρα τους ε, πουλάμε την εσωτερική αγορά και ο κύριος Κάμερον ε, και κάποιοι άλλοι και ο κύριος Μόντι φυσικά έγραψαν μια επιστολή σχετικά με τις αρετές της εσωτερικής αγοράς και όλη αυτή τη δυναμική δεν τη βλέπουμε σε αυτές τις 20 προτάσεις. Εάν λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτές τις 20 προτάσεις, τότε να προσθέσουμε ότι είναι 20 προτάσεις ε, στο πλαίσιο της ιστορικής αγοράς. Αν θέλουμε να έχουμε κάποια δραστηριότητα στο εξωτερικό και στην περίπτωση αυτή χρειάζεται τουλάχιστον να αναφέρουμε το ζήτημα της δυνατότητας μεταφοράς των ε, συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και θέλουμε να έχουμε μια ευρύτερη, μια σφαιρικότερη προσέγγιση. ένα πολίτη ή μια επιχείρηση ε, στην εσωτερική αγορά τι ζητήματα αντιμετωπίζει και τον προβληματίζουν. Έχουμε άλλα θέματα που μας απασχολούν και μέσω τροπολογιών, τίποτα δεν μας απαγορεύει να θίξουμε αυτά τα θέματα που η Κομισιόν δεν τα έχει συμπεριλάβει στις 20 ε, ανησυχίες. Ε, λοιπόν, εγώ έχω ένα ζήτημα που, για το οποίο θα καρθούσε και τροπολογία και αφορά και εργασίε τη Επιτροπή μα στο παρελθόν, πρόκειται για το ζήτημα της κοινωνικής στέγασης και των ε, αστέγων. Είναι θέμα του, το θέμα του ανταγωνισμού και των κρατικών επιδοτήσεων είναι ζητήματα ύψης της σημασίας και δεν ε, αναφέρονται στις 20 αυτές προτάσεις της Κομισιόν. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτά είναι δύο ζητήματα που πρέπει να πάμε, για τα οποία πρέπει να πάμε παραπέρα. Κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορείτε να κάνετε εσείς ε, ως συγγύδρια μέσα στο γνωμοδότησή σας, αλλά ε, οι τροπολογίες θα μας το επιτρέψουν. Έχετε τον λόγο κυρία Συγγύδρια για να κλείσουμε τη συζήτηση. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Η Γιούτα Στάνιζουκ ανέφερε κάτι το σημαντικό, πράγματι. Είναι δύσκολο τα σημεία αυτά τα οποία αναφέρονται στην, ε, στην ανακοίνωση της Κομισιόν ε, δεν έχουν κάποια πρόταση επίλυσης. Ε, δεν είναι ικανοποιητική αυτή η κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή. Γι' αυτό ακριβώς η δική μας η δουλειά ως Επιτροπή Απασχόλησης είναι να συνεισφέρουμε ιδέες ας μην είναι και πάρα πολύ λεπτομερείς απλά να πούμε ποια κατεύθυνση θέλουμε εμείς να ακολουθήσουμε ως ε, Ευρωκοινοβούλιο και οπωσδήποτε και αυτά τα θέματα ε, ταιριάζουν εδώ πέρα και οι δημόσιες προμήθειες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα πρέπει νομίζω να βάλουμε σχετικές τροπολογίες. Είμαι ανοιχτή σε αυτό. Αλλά επίσης θεωρώ πως θα πρέπει να συνεισφέρουμε και κάποιες ιδέες. Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης είναι μια δυσκολία όχι μόνο η μεταφορά των δικαιωμάτων και ο υπολογισμός τους, αλλά στα συστήματα τα ίδια, π.χ. τα συνταξιοδοτικά. Εάν κάποιος δουλεύει ε, part-time, παραδείγματο χάρη, έχει αυτομάτως ένα μειονέκτημα, κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται. Είμαστε σε μια ε, εσωτερική αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Και αυτό είναι νομίζω αυτό το οποίο πρέπει να διευκρινίσουμε εμείς. Θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε όταν εξετάσουμε την έκθεση κυρία για τον ε, κοινωνικό αποκλεισμό. Ωραία. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτό το σημείο και το χρονοδιάγραμμα προβλέπει να υποβληθούν οι τροπολογίες για το σχέδιο αυτό μέχρι τις 6 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι. Θα τις εξετάσουμε 26-27 Μάρτιου και θα ψηφίσουμε από αυτού 23-24 Απριλίου. Η Επιτροπή ΙΜΚΟ θα πρέπει να εκφραστεί στην έκθεση της κυρίας Βαστός στις 19 Ιουνίου. Τελειώσαμε τώρα αυτό το σημείο της σημερινής διάταξης και περνάμε στην... στις ψηφοφορίες. Στο σημείο 9, έκθεση της κυρίας Μωρά. Για την υγεία και ασφάλεια στον τόπο εργασίας στην, σε εργαζόμενους που εκτίθενται σε κινδύνους που φυσικού φυσικούς παράγοντες, λαμβανικά παιδεία κυρίως, δεν πρόκειται για την οδηγία εξουσίας, αλλά εκείνη που έχει σαν στόχο να παρατείνει την ισχύουσα. Άρθρο 1. Τροπολογία 2. Καρή Μαντελή, Ελίζα και άλλων. Ταυτόσιμο με την τρία της κυρίας Ράπτη. Ψηφίζουμε και τις δύο αυτές τροπολογίες. Η εισηγήτρια είναι κατά των δύο τροπολογιών. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του σχεδίου έκθεσης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μία ψήφος κατά, μία αποχή. Και ψηφίζουμε την πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Με την ίδια πλειοψηφία. Εγκρίνεται και συγχαίρουμε την εισηγήτριά μας. Α, όχι, όχι, για ένα λεπτό. Πολύ βιάζομαι. Όπως ξέρετε, βάσει της που μόλις έγινε, θα άνοιξει διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο, στην οποία θα βρισκόμαστε σε διαδικασία συναπόφασης. Και λόγω του κατεπήγοντος, θέλουμε και εκατόμιση εντολής που ορίστη, να καταλήξουμε σε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Βάσει του άρθρου 70 και του παρατήματος 21 του, 21 του κανονισμού μας, θα πρέπει να ελέγξω, με τη βοήθειά σας, τη σύνθεση της ομάδας διαπραγμάτευσης, τη φύση της εντολής και να σας ενημερώσω για το, το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων. Προτείνω λοιπόν η ομάδα διαπραγματεύσεων να αποτελείται από την εισηγήτρια, τους σκιώδες συζητητές και να είμαι πρόεδρος αντιπροσωπείας αυτής. Δεν διαφωνεί κανένας. Ωραία, θαυμάσια. Όσον αφορά για την εντολή των διαπραγματεύσεων θα είναι βάσει αυτών που αποφασίσαμε αυτή τη στιγμή. Συμφωνούμε όλοι, θαυμάσια. Θα ήθελα να σας ε, ενημερώσω ότι ο πρώτος ημέρας διάλογος με το Συμβούλιο και το Κομισιόν προβλέπεται για τις 5 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα. Προς επιβεβαίωση. Αν δεν διαφωνεί κανένα, σα ευχαριστώ και θα σας ε, παρουσιάσουμε σε επόμενη συνεδρίαση την πρόοδο των εργασιών. Σημείο 10. Έκθεση Μιλάν Κάρμπονοχ για την του κανονισμού για του συνοσμό των συστημάτων κοινωνική ασφάλεια και τον κανονισμό καθορισμό τη ε, διαδικασία εφαρμογή του κανονισμού. Άρθρο 1, σημείο 1. Νέο. Τροπολογία 14 του εισηγητή. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 1, ε, σημείο 1, άρθρο 9, 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1, 2, α, 16 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1-4, τροπολογία 2 του εισηγητή με μια προφορική τροπολογία που πρόκειται για μια γλωσσική διόρθωση. Όλη η τροπολογία είναι... Α, όχι, όχι. Λοιπόν, πρέπει να βοηθήσουμε την τροπολογία με μια ε, διόρθωση γλωσσική. Ψηφίζουμε τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 3, σημείο 4. Β, Ι, Ι, Τροπολογία 3 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 και 22 ταυτόσημες ψηφίζουμε από κοινού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 23 και 24. Υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνονται. 5 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 6 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 26 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 28 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 31 με μια τροπολογία γλωσσική, δεν διαφωνεί κανένα για τη γλωσσική τροπολογία φαντάζομαι, υπέρ της 31 κατά αποχές εγκρίνεται. 32 το εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται. 33 το εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται. 8 το εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται. 9 το εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται. 34 της κυρίας Ουμεν Ρόιτν. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές απορρίπτεται. σκέψη 4. Η 10 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχή. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 10. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τιολογική σκέψη 5. Τροπολογία 11 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο της ε, πρότασης ως τροποποιήθηκε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ, είναι κάποιος που δεν έχει την κάρτα του μαζί. Άρχιε ψηφοφορία. Του le πιβωτή ψηφοφορία. 42 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται η πρόταση αυτή και περνάμε στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Tout le monde a pu Ψήφισαν όλοι υπέρ της ψηφοφορίας. 42 υπέρ, καμία ψήφος κατά και μία α... αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Αυτό σημαίνει ότι με το κείμενο σύμφωνα και με το Συμβούλιο και μπορούμε να το εγκρίνουμε λοιπόν οριστικά στην επόμενη Σύνοδο Ολομελίας. Θέλετε κάτι για διαδικαστικό να αναφέρετε παρακαλώ. Ναι, μια παρατήρηση, κυρία Πρόεδρε. Στη διάρκεια της ε, ψηφοφορία παρατήρησα πως 75% των ψηφοφοριών δεν κοιτάτε καν. Ε, μια και μας βλέπουν στο διαδίκτυο, καλό είναι να τηρούμε και τα προσχήματα. Στα τρία τέταρτα δεν, δεν κοιτάξτε καν ποιο σήκωνε το χέρι. Είναι γνωστή αυτή η παρατήρηση της ομάδας σας, δεν ξέρω γιατί το είχα κατά νου πάντως στις ε, ψηφοφορίες. Θυμάμαι που το, το είχε θίξει η ομάδα σας. Μα, μα γι' αυτό σας λέω ομάδα. Και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ήξερα πως δεν χρειαζόταν να κοιτάω κάθε φορά γιατί η πλειοψηφία ήταν συντριπτική υπέρ του. Οπότε δεν να Κάνω όλη τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Και οπωσδήποτε υπάρχει η δυνατότητα τελική ψηφοφορία να γίνει ηλεκτρονικός. Οπότε απορρίπτεται η παρατήρησή σας. Περνάμε τώρα στο σημείο 11 για το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών και την γνωμοδότηση της κυρίας Σούμπερ άρθρο 2.1 73 σύπελ. Υπέρ, κατά, για να ελέγξουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. 18 υπέρ, 24 κατά και μία αποχή. Απορρίπτεται 73. 74 του κύριου Μπέκερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 75. Είναι συμβατή υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 2 παράγραφος 2. Ταύλα 2. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 2 παραγραφός 2 με ένα νέο 2α. Συμβαστική τροπολογία β. Υπέρ. Κατά. Συγγνώμη, 78 του κ. Μπουλό. Συγγνώμη, η 78 του κ. Μπουλό ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 16 κατά, 3 αποχές. Εγκρίνεται, σαφέστατα. 2, παράγραφος 2, Παύλα 3, συμβαστική τροπολογία Β, από 5 πολιτικές ομάδες. Όταν ψηφίσουν μία γραμμή θα περιοριστεί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 2, παράγραφος 2, 3, νέο βάσει της τροπολογίας 13 ε, τη συζητήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 3 παράγραφος 1α νέο. Τροπολογία 82 του κυρίου Μπουλό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 3 παράγραφος 1 παύλα 1 συμβαστική γάμα από 5 ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 3 παράγραφος 1 παύλα 2. 86 του κυρίου Μπουλό υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 κιόντς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αυτό 3 παραγραφός 1 παύλα 3 τροπολογία 14 της συζυγήτριας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 κιόντς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 3 παράγραφος 1 παύλα 3α Τροπολογία 89 Τσούβερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρθρωτία παράγραφος 1 Παύλο 5. Παύλα 5, συμβαστική δέλτα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 3, παραγραφός 1, 5α νέα, τροπολογία 92 τη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Η 93. Ελέγξουμε την 93. Άχι ψηφορία, πέρες ψηφορίες. 20 υπέρ, 20 κατά. Α, απορρίπτεται. Ήταν χρήσιμος ο έλεγχος λοιπόν. 94. Πέκερ, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 95 με μια προφορική τροπολογία, δεν διαφορεί κανένα με προφορική τροπολογία, ψηφίζεται υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 96 του 2 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 97 μπουλό υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 98 μπουλό υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 99 μπουλό υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 100 σιπέλ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 μπέκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 λομπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 λομπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 μπέκερ υπέρ να ελέγξουμε την 103 να την ελέγξουμε. Ευχαριστώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. 21 υπέρ, 21 κατά. Η ίδια κατάσταση όπως προηγουμένως. 104. Ναι, σας μέτρησα εσάς. 21 υπέρ και 21 κατά. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία υπέρ. Προσθέσουμε τη δική σας ψήφο και τη δική μου και δεν εγκρίνεται άμα είναι ισοψηφία. Είναι η μόνη μας κανόνας αυτός ε, του κοινοβουλίου. Παρεμβάσει εκτός μικροφώνου. Deux socialistes qui sont mauvais élèves de la carte. Οι δύο σοσιαλιστές ε, δεν είναι καλοί μαθητές. Η πρόεδρός σας και ο κύριος Σόλε. Δεν έχουν δηλαδή την κάρτα μαζί τους. Α, παρδού! Α, Παρεμβάσει εκτός μικροφώνου. Δεν γίνεται, λέει η πρόεδρος. Δεν γίνεται. 23 υπέρ λοιπόν και 19 κατά. Αλλά η τροπολογία Λόμπερ εγκρίνεται. Με συγχωρείτε και σας ευχαριστώ κύριε Λέ που επαγρυπνείτε. 104 Μπέκερ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 105 Σίπελ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τη λογική σκέψη 1, 16 σε δύο τμήματα. το σύνολο της τροπολογίας χωρίς εμφασίζοντας στην εθνότητα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτός ο, ε, ο τύπος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ετολογία 1 α νέα, τροπολογία 1 τσούβερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 Παπαδοπούλου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται. 18 σύπελ υπέρ κατά εγκρίνεται. 19 σύπελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική σκέψη 3 συμβαστική ε, 5 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4. Τροπολογία 22 Κιόντς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εθελώς και 4 4α, νέα. Τροπολογία 23, Παπαπαπούλου, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 24, Μπέκερ, υπέρ, κατά, αποχές. Για να ελέγξουμε την 24, Μπέκερ. Ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίες. 28 υπέρ, 15 κατά. Εγκρίνεται σαφέστατα. 25 συμβατή υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26 Ρέγνερ υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 3 Τσούμπερ υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 27 Παπαδοπούλου υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται αιτιολογική 7, τροπολογία Και αν τη κανένα, θα έλεγα να αντιστρέψουμε τη σειρά τη ψηφοφορία. Γιατί αν υπάρχει ένα συμβασμό πάνω σε ένα κείμενο, πρέπει να ψηφιστεί πρώτα η συμβαστική τροπολογία. Συμφωνείτε όλοι. Ωραία. Λοιπόν, συμβαστική F5 πολιτικών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Με συγχωρείτε που κάνω αυτή την παρατήρηση κατά τη διάρκεια τη ψηφοφορία, αλλά κάτι δεν με, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε μία, ε, ψηφο, μία τροπολογία πριν από τη συμβαστική, εκτός αν πρόκειται η διαγραφή του κειμένου. Ε, Τριολογική σκέψη 7. 2035 35 σύπελ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τριολογική σκέψη 8. Η ίδια κατάσταση όπως για την 7. Αλλά έχει αποσυρθεί βέβαια η άλλη τροπολογία. Ε, συμβαστική Ζ, υπέρ, κατά αποχέ. εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 9, συμβαστική Ι, πέντε πολιτικών ομάδων, υπέρ, κατά απόχέ. εγκρίνεται. C'est un nouveau paragraphe. Ah ouais, donc c'est deux parties du paragraphe. Donc, euh, toujours sur le considérant. Στην ίδια τελική σκέψη 9, δεύτερη συμβαστική τροπολογία H, α, ήτα, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Μετά περνάμε στη 47 τσούβερ 9α νέο, υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. 48 ΣΥΠΕΛ σε δύο τμήματα. Το σύνολο του κείμενου χωρίσκει. Αυτό που έχει δεχθεί κατά μέρο υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται το υπόλοιπο του κειμένου υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. Τουλική σκέψη 10. 49 κόντ υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 50 λομπέρ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 7 της ηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ετιολογική σκέψη 11. Συμβαστική ζή Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική 12. Τροπολογία 9 της ηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 πουπάκες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 καταπίπτει και περνάμε στην 55 μπουλό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Μητολική σύμφη 13 σε δύο τμήματα Συμβαστική κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική L το δεύτερο τμήμα του αιτιολογικής σκέψη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά έχουμε την τροπολογία 10 τσούμπερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 πλάμπ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 βουλό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 ρέγνερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, το 15 τροπολογία 66 μπέκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Φιλική 17, τροπολογία 67 μπέκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Του λυγής 18, τροπολογία 68, σύπερ σε δύο τμήματα. Πρώτα, το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το υπόλοιπο του κειμένου υπέρ, κατά αποχές απερίπτεται. Α, δεν χρειάζεται. 69 σύπερ, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 λιπέρ, υπέρ mm. κατά αποχές εγκρίνεται 71 μπέκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 στους 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο της γνωμοδότησης ηλεκτρονική ψηφοφορία Άρη η ζωφορία. Πέρασε η ζωφορία. 38 υπέρ, δύο εποχές, 2 κατά και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια αντιπρόεδρο για την πρώτη έκταση. Κύριε Ρή. Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στο σημείο 28 που ψηφίσαμε. Για το 28 λέω. Ψηφίσαμε, αλλά ομολογώ ότι δεν ήμουν πολύ ικανοποιημένο με τη σειρά με την οποία ψηφίσαμε. Γιατί συνήθως εάν μια τροπολογία τροποποιούσε σημαντικά τον συμβιβασμό, Ψηφίσαμε πρώτα την άλλη τροπολογία και μετά το, τη συμβαστική. Δεν είναι δηλαδή γενικό κανόνα αυτό θα πρέπει η τροπολογία να ψηφιστεί πριν από την συμβαστική. Αν δεν είναι πολύ σημαντικό το θέμα, από την άλλη μεριά θα πρέπει η γραμματεία όταν προετοιμάζει τον κατάλογο της ψηφοφορίας να το κάνει έγκαιρα, όχι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας να έχουμε νέες ερμηνείες. Θα πρέπει να διευκρινιστεί. Υπάρχει αυτός ο κανόνας ότι αν πρόκειται να τροποποιηθεί ένας μια συμβαστική τροπολογία σημαντικά από μια άλλη τροπολογία θα πρέπει να γίνει ψηφοφορία πριν από τη εκείνη τη συμβαστική. Ο κύριο Σέρκα. Πρόεδρε, πιστεύω ότι υπάρχει παράδοση στην Επιτροπή μας όπως ε, είπατε και εσείς, όταν υπάρχει συμβαστική τροπολογία τότε οι ατομικές τροπολογίες πρέπει να έπονται. Αυτή είναι μια πρακτική. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ε, προσεκτικοί όταν ε, ψηφίζουμε, αλλά τα καλά στοιχεία θα πρέπει πάντα να τα διατηρούμε. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, η έννοια μιας συμβαστικής τροπολογίας είναι να κινητοποιηθούν ο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ε, των συναδέλφων για να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η παράδοση προβλέπει ότι πρώτα ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία. Βλέπω κύριε ότι εσείς ε, θέσατε το σημείο αυτό μετά την ψηφοφορία. Άρα φαντάζομαι δεν ήταν αποφασιστικό το σημείο για σας. Και άμα διαβάσετε το άρθρο 160 παράγραφο 4 του κανονισμού βλέπετε τι λέει. Είναι το άρθρο για τη βάση ψηφοφορίας. Η πρόεδρος μπορεί επίσης να προτείνει συμβαστικές τροπολογίες βάσει της παραγράφου 4 και αν υπάρχει συμβαστική τροπολογία αυτή ψηφίζεται κατά προτεραιότητα. Προτεραιότητα. Και νομίζω αυτό το κανόνα εφέμωσα. Κύριε Ρία, έχετε το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ δεν θέλω να τροποποιηθεί η ψηφοφορία τώρα. Δέχομαι ότι έτσι ψηφίσαμε, αλλά θα ήθελα οι κανόνες να είναι ξεκάθαροι έχουμε εισακάγει κάποια παράδοση ότι κατά κανόνα ψηφίζουμε κατά προτεραιότητα πρώτα συμβαστικέ τροπολογίε σε γενικέ γραμμέ. Μπορώ να συμφωνήσω. Αλλά εδώ στην Επιτροπή μα είχαμε την ε, παράδοση ότι μια συμβαστική τροπολογία ε, τροποποιείται σημαντικά ε, πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα αυτή την τροποποιητική, αν θέλετε, τροπολογία επί της συμβαστικής. Κοιτάξτε, δεν θα ε, παρατείνουμε τη συζήτηση αυτή εν μέσω της πληροφορίας. Αν θέλετε να το ξαναθίξετε το θέμα αυτό, μπορούμε να το κάνουμε στην συνεδρία των συντονιστών. Εκεί είναι ε, το σωστό να το κάνουμε. Αλλά σας παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά το άρθρο 160 του κανονισμού του σώματος. Με προσοχή είναι ένας ε, κανόνας που επιβάλλεται στις ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές βάσει ενός άρθρου, όπως είπαμε του κανονισμού μας. Περνάμε τώρα στο σημείο 12 της ημερησίας μας διάραξης. Αναγνώση και πρόσθεση διασυνορικών εθελοντικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει η έκθεση γνωμοδότης κυρίας Άρκιν, παράγραφος 1. Συμβαστική τροπολογία καταρχήν. Συμβαστική α, που έχουν υποβληθεί από διάφορους ε, βουλευτές. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά περνάμε στην τροπολογία 6 που θα ψηφίσουμε αργότερα μέσα στην τροπολογία G. <clears throat> Για την παράγραφο 1α νέα συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επίσης, τροπολογία F, συμβαστική τροπολογία F. Υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Πέραφος 2, συμβαστική σε, γάμα, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 2α νέα, τροπολογία συμβαστική δέλτα, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Νέο σημείο βάση τροπολογίας 23 ε, της κυρίας Ρουτσολή καταπίπτει. Ψηφίζουμε λέμε λοιπόν την 24. Πληγεβιτσιούτα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 της ίδιας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στην παράγραφο 3 μία πρόταση διαγραφής του κυρίου Χέλμερ, που είναι η πρώτη που θα ψηφίσουμε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά περνάμε στην τροπολογία 32 Ροντσούλη με μια προφορική τροπολογία της ίδιας. Δεν διαφωνεί κανένας. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 36, Ροντσούλη, που τους ίδιους υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 37, Λαμπέρ, υπέρ, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Συμβαστική Ζ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στην παράγραφο 6, συμβαστική άσχη. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά, τροπολογία 47 ραντσούλη υπέρ κατά. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ τη 47 κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 54 πλάμ υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 55 ροντσόλι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Άμε με συγχωρείτε. Στην παράγραφο 7 δεν ψηφίσαμε τροπολογία Ιώτα. Υπέρ της τροπολογίας Ιώτα. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Συμβασική G. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60 πλάμπ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 σάγια υπέρ κατά για να ελέγξουμε. Την 61, τροπολογία 61. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 22 κατά. Απορρίπτεται. 18 υπέρ, 24 κατά. Εντάξει, απορρίπτεται πάντως. 62 κόντς υπέρ. Κατά. 62 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 63 άρκιν υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 Χέλμερ σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα κατά αποχές απορρίπτεται οπότε δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε δεύτερο τμήμα τροπολογία 66 Χέλμερ καταπίπτει Σύνολο του κείμενου αστροποποιήθηκε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Α, ο κύριο Μακαμλόκ. Με συγχωρείτε. Δεν ψηφίσαμε τις 43. Μα υπερψηφίσαμε τη συμβαστική ήττα. Λοιπόν, ψηφίσουμε τώρα το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικά. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ψήφισαν όλοι υπέρ της ψηφοφορίας. 39 υπέρ, μία ψήφος κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Euh, Τελειώσαμε λοιπόν την ε, ηλεκτρονική αυτή ψηφοφορία και περνάμε στην αλληλεγγύη απόψεων μέσα στα πλαίσια της έκθεσης κυρία Σάρκιν για το Ευρωπαϊκό Τομείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Συνάδελφοι, να σας ζητήσω να επιστρέψετε στις θέσεις σας, διότι ο χρόνος τρέχει. Σημείο 13. Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση για την περίοδο 2014-2020. Έχουμε ακρόαση, ανταλλαγή απόψεων, και προτείνω να δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Άρκιν. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συζητάμε σήμερα νέες προτάσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, αλλά πρέπει να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτό υπάρχει ένα ζήτημα που μας απασχολεί. Η απόφαση του Συμβουλίου πέρσι να μην συνεχίσει με την παρέκκληση της κρίσης και η ΕΟΚΕ εξέφρασε την ε, κατάπληξή της και η Επιτροπή των Περιφερειών επίσης και βέβαια ξέρουμε και την άποψη του Κοινοβουλίου. Απλά στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης νομίζω πως τίθενται σημαντικά ζητήματα για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής. Επίσης πρέπει να διδαχτούμε από την μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής. Κάποια από τα ζητήματα που τέθηκαν μέχρι στιγμής, έτσι σύντομα, το να δρα, ε, το Ταμείο, αλλά βεβαίως ε, εδώ πέρα έχουν ευθύνη και τα κράτη-μέλη. Μπορούν να εφαρμόζουν τα μέσα με την υποβολή της αίτησης. Ε, το ποσοστό συγχρηματοδότησης, πρόβλημα σε κάποιες χώρες, το όριο, το κατόφλι για τον αριθμό εργατών και επίσης όλο και περισσότερα κράτη-μέλη υποβάλλουν αιτήσει, αλλά όχι όλα. Ένα άλλο ζήτημα, συμπερίληψη των κοινωνικών εταίρων και συνέργεια με τα λοιπά ταμεία, το κοινωνικό κτλ. Η πρόταση η ίδια τώρα έχει στόχο να δίνει άπαξ στήριξη σε εργαζόμενους που έχουν χάσει τη δουλειά τους σε διάφορους τομείς. Και οι όροι είναι μεταφορά της βιομηχανίας σε τρίτες χώρες, μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές λόγω της παγκοσμιοποίησης και βεβαίως ε, η επίδραση στην τοπική και περιφερική οικονομία των απολύσεων. Υπάρχουν νέες προτάσεις. Απολύονται οι εργαζόμενοι επίσης ε, αποτέλεσμα, ως αποτέλεσμα αναπάντεχης κρίσης, νέα πρόταση. Επίσης, το βασικό σημείο συζήτησης, η συμπερίληψη των αγροτών. Και σημειώνουμε πως την ε, γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ ήταν κατά. Και η Επιτροπή των Περιφερειών πρότεινε πως πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή και βεβαίω θα αλλάξει έτσι η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε τώρα υπάρχουν δύο διαφορετικά ταμεία τέτοια. Επίσης και το εάν μπορούν να συμπεριληφθούν και οι οικογένειες των αγροτών. Επίσης για πρώτη φορά περιλαμβάνει και προσωρινούς ε, εργαζόμενους καθώς και ιδιοκτήτες ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα μείνω σε αυτά έχει και άλλα πολλά. Θα ήθελα να μάθω τι έχουν να πούν οι συναδελφοί μας. Και ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω στο τέλος. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Λόγω του κυκλοφοριακού χάους των Βρυξελών θα πρέπει να αντιστρέψουμε στις ε, παρουσιάσεις των εμπειρογνωμόνων Προτείνω σε τούτου να ξεκινήσουμε τον δεύτερο εμπειρογνώμονα, κύριο Κάρλος Τορτουέρο Μαρτίν, αναπληρωτή διευθυντή στο Υπουργείο Εργασίας και Μετανάστευσης στην Ισπανία. Έχετε το λόγο για δέκα λεπτά. Κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, καταρχήν ε, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας ε, έγινε για να σας ε, μιλήσουμε για την εμπειρία στην Ισπανία Ειδικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής το 2010-2011 λειτουργήσε το Ταμείο, μάλλον το 2008 λειτουργήσε και εποφελθήκαμε από αυτό το Ταμείο στηρίζοντας 18 προγράμματα, 18 σχέδια. τα οποία αφορούσαν περίπου 10.000 εργαζόμενους οι οποίοι μπόρεσαν να αναδιοργανώσουν την ζωή τους, να βελτιώσουν τις ικανότητές τους, την κατάρτισή τους για να αποκτήσουν μια, νέες δυνατότητες απασχολησιμότητας τη στιγμή αυτή που διανύουμε μια πολύ σκληρή κρίση οικονομική και κρίση στον τομέα της απασχόλησης. Τώρα τα 18 προγράμματα λοιπόν, 5 αφορούσαν ε, το παγκοσμιοποίηση και 13 αφορούσαν το κεφάλαιο οικονομική κρίση. Δηλαδή, ε, η τροπολογία η οποία εισήχθη για να στηρίξουμε αυτή την οικονομική κρίση μέσω του Ταμείου. Τώρα, σε ό,τι φορά τα κριτήρια παρέμβασης, να πω ότι ένα πρόγραμμα αφορούσε την στήριξη μιας επιχείρησης 1.300 εργαζομένων, 26 προγράμματα αφορούσαν το άρθρο 2 του κανονισμού, δηλαδή ε, τομεακή κρίση, και μόνο ένα πρόγραμμα αφορούσε το άρθρο C, που τις υποβαθμισμένες ε, ζώνες ε, όπου η ανεργία ξεπερνούσε το 10%. Τώρα, σε ό,τι φορά τους οικονομικού κλάδου, τέσσερα προγράμματα αφορούσαν ε, στον τομέα των αυτοκινητομηχανίας, ε, τρία στην εφαντουργία, δύο στον κατασκευαστικό τομέα, δύο προγράμματα ε, στην κατασκευή θυρών, ένα τομέα στην κεραμική, ένα πρόγραμμα στο το μέρο μαρμάρων, ένα στο εμπόριο και ένα στο ότι φορά την ε, αθλητική υπόδηση. Τώρα, όπως είπα, 10.000 άτομα τα οποία έλαβαν άμεση στήριξη από το Ταμείο και το 32% ήταν γυναίκες και το 67,9% ήταν άνδρες. Το ποσό της βοήθειας είναι 41 70.000 ε, μάλλον ανά πρόσωπο η στήριξη ήταν 4.239 ευρώ, δηλαδή κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που αυτή τη στιγμή ήταν τη τάξη του 4.680 ευρώ. Να πω επίσης ε, πως σύμφωνα με την εμπειρία που αποκτήσαμε αυτή την περίοδο ε, τη σημασία που έχει το συγκεκριμένο ταμείο. Το ταμείο αυτό προσπαθεί να επιτύχει μια εντατική συνεργασία ανάμεσα στους εμπλεκομένους ε, συνεργασία σε εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό, τοπικό και ιδιαίτερα μέσω της συμμετοχής ε, επιχειρηματιών αλλά και προσώπων των εργαζομένων. Είναι μια εμπειρία η οποία καταδεικνύει τις προσπάθειες των ενδιαφερομένων προκειμένου να επιληθούν τα προβλήματα τα οποία οδηγούν σε απώλειες θέσεις εργασίας στον, στον οικονομικό τομέα. Να πω επίσης ε, τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που έχει το πρόγραμμα. Αυτό το ταμείο λοιπόν αφορά σε συγκεκριμένα μέτρα που εστιάζονται στο πρόσωπα, στις ανάγκες τους και ειδικά παρέχει ευελιξία και προσαρμοστικότητα την στιγμή εφαρμογής βελτιώνει την απασχολησιμότητα διότι βελτιώνει την, τα προσόντα των προσώπων. Να πούμε ότι η χώρα μας με τα προγράμματα του Ταμείου Προσαρμογής και το δείκτες ε, επανέβρεσης εργασίας φτάνει σε υψηλά ποσοστά τη στιγμή που ε, διανύουμε οικονομική κρίση και είναι προφανές ότι βελτιώνει τη δυνατότητα απασχολησιμότητα ε, και η ικανότητα των ε, προσώπων να μεταφερθούν και να βρουν απασχόληση σε άλλους κλάδους. Όπως είπα, δημιουργούμε συνέργειες μεταξύ των εμπλεκομένων και υπάρχει ένας πολύ ψηλό βαθμός εγκύτητας και ε, οι συστάσει που θέλουμε να κάνουμε για την προσεχή περίοδο είναι εξή. Να συνεχιστεί η περιφερειακή αυτή εφαρμογή του Ταμείου, να συνεχίσουμε με την σημασία που έχει η διατήρηση αυτού του Ταμείου. Κατά την άποψή μα είναι πολύ σημαντικό το, η, κρίση ε, να μπορέσει να μας οδηγήσει σε μια καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος. Υπάρχουν λοιπόν ε, ε, δημοσιονομικές ε, περικοπές και θεωρούμε ότι η συγχρηματοδότηση που αφορά τα έτη 2009-2001 και αν έρχεται στο 75% είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να φροντίσουμε να διατηρήσουμε. Οι αυτόνομες κοινότητες στην Ισπανία αντιμετωπίζουν δυσκολίες για να πέσει αυτό το ποστό στο 50%. Ε, θα πρέπει λοιπόν η κοινωτική στήριξη να διατηρήσει την σημασία της ε, κατά την άποψή λοιπόν. Θα ήταν ιδιαίτερα θετικό να προσπαθήσουμε να, να θεωρήσουμε τον αριθμό των ε, εμπλεκομένων εργαζομένων. Ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ενδεχόμενες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. ορίζω και τον τρίτο πυρογνώμονά μας. Ε, θα του επιτρέψω να πάρει μια ανάσα και να ακούσει τις ε, τη συζήτησή μας. Δίνω το λόγο στην κυρία Μακεβιλιεύσκη, συγγνώμη για την προφορά, διευθύντρια στο Υπουργείο εργασία ε, τη Λιθουανία. Συγγνώμη που σκότωσα το όνομά σα προφέροντα το. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ. Ε, προσωπικά Χαίρομαι για το ότι η κυρία Λιγκεβιτσούτα, η πρώην υπουργό μου πέρα, μπορεί να προφέρει το όνομά μου. Μην ανησυχείτε, πάντα όλοι οι αλλοδαποί δεν μπορούν να προφέρουν το όνομά μου. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι εδώ πέρα σε διαφορετική επιτροπή για να παρουσιάσω την εμπειρία μας για το Ταμείο της παγκοσμιοποίηση στη Λιθουανία. Έχουμε αρκετή εμπειρία γιατί ξεκινήσαμε ευθύ εξ αρχής με το Ταμείο αυτό για να εκμεταλλευτώ το χρόνο που έχω. Να σας αναφέρω λοιπόν ποιες ήταν οι εμπειρίες μας. Και να προτείνω μετά α, ε, κάποια πράγματα για το νέο κανονισμό 2014-2020. Στη Λιθουανία η διαχειριστική αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου στην ε, προσαρμογή είναι το Υπουργείο μας και οι υπόλοιπες αρχές που εμπλέκονται είναι το Υπουργείο Οικονομικών που ασχολείται με τα ζητήματα ε, με το να κρίνει ε, το εάν ε, μια συγκεκριμένη εταιρεία ή κλάδος έχει υποστεί τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, οπότε οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται μόνο από το δικό μας Υπουργείο, αλλά και από το Υπουργείο Οικονομικών και βεβαίω από ένα τριμερές συμβούλιο με τους κοινωνικούς εταίρους που συμμετέχουν ε, ενεργά στη συζήτηση. Συζητήσαμε όταν συζητάμε τη δυνατότητα χρήσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Να επισημάνω επίσης πως οι κοινωνικοί εταίροι δεν συμμετέχουν στη χρήση των ε, κονδυλίων αυτών. Επίσης, η Λιθουανία έχει εφαρμόσει πέντε έργα από το ταμείο αυτό. Πρέπει να σημειώσω εδώ πέρα πως ε, είχαμε την ευκαιρία ένα από τα πρώτα έργα τα οποία εφαρμόσαμε ήταν ε, όταν απολύθηκαν οι εργαζόμενοι μιας ε, υφαντουργίας. Μια άλλη περίπτωση ήταν πάλι απολύσεις από μια εταιρεία ε, που χρησιμοποίησαμε τον αναθεωρημένο κανονισμό τα άλλα έργα ήταν τομεακές εφαρμογές και εδώ πέρα θα ήθελα να σημειώσω πως και τα πέντε έργα εφαρμόστηκαν. Επιτυχώς συμπληρώθηκαν και είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Όχι βέβαια τα ίδια σε όλα τα έργα. Στα τρία τελευταία έργα διευκολυνθήκαμε από το ότι Σύμφωνα με την ΝΑΤΣ 2 η Λιθουανία είναι μία περιφέρεια και τα έργα παρουσιάστηκαν ε, για λογαριασμό της χώρας. Τα καλύτερα αποτελέσματα τα είχαμε στην εφαρμογή των έργων που είχαν να κάνουν με τις ε, απολύσεις ατόμων σε μεμονωμένες εταιρείες. Σε γενικές γραμμές όμως καταφέραμε να χρησιμοποιήσουμε και να ε, εμπλακούν γύρω στο 90% των συμμετεχόντων και χρησιμοποίησαμε γύρω στο 70% των διαθέσιμων κονδυλίων. Το καλύτερο αποτέλεσμα το επιτύχαμε στο πρώτο έργο σε μια εταιρεία ε, στην υφαντουργία που ανέφερα Μιλάμε για ένα 99% ε, απορρόφησης των κονδυλίων. Τα, στα άλλα έργα ήμασταν γύρω στο 69%. Όσον αφορά τώρα την περίοδο εφαρμογής, είχαμε ένα επίπεδο νέας απασχόλησης γύρω στο 63% είτε μόνιμη είτε προσωρινή εργασία. και όπως ε, προβλέπει ο κανονισμός χρησιμοποιήσαμε ενεργά μέτρα τα οποία είναι ε, προβλέπει η νομοθεσία μας για τη στήριξη της απασχόλησης και η κυβέρνηση επίσης έλαβε και επιπλέον μέτρα για τους ανθρώπους οι οποίοι απολύθηκαν. Κάποια από αυτά τα μέτρα ήταν επιτυχή και ε, μεταφέρθηκαν και στον νόμο περί στήριξης της απασχόλησης. Βεβαίως, βλέπετε εδώ πέρα, παραδείγματα, κάποια από τα οποία περιγράφονται στην ε, ανακοίνωση της Κομισιόν διοργανώσαμε αρκετά συνέδρια όπου προσκαλέσαμε τους συμμετέχοντες να μας μιλήσουν για τις επιχειρήσεις τους. Η εμπειρία μας όμως είναι... έχει δύο πτυχές. Βεβαίως το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση είναι συγκεκριμένο, στοχευμένο και βασίζεται στις ε, συγκεκριμένες ανάγκες απολυμένων εργαζομένων για να μπορέσουν να ξαναβρούν δουλειά και να προετοιμαστούν για κάποιες ε, θέσεις εργασίας. Η θετική εμπειρία λοιπόν από την διαδικασία αίτησης είναι η αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης στο 65% το δεκατόφλι μειώθηκε στους 500 απολυμμένους και βεβαίως ξέχασα να αναφέρω ε, για μία περίπτωση είχε ως αιτία την παγκοσμιοποίηση, οι άλλες ε, είχαν την οικονομική κρίση. Αλλά και πάλι είχαμε στήριξη από το Ταμείο. Όλα τα, τα μέτρα βεβαίω ε, τα εφαρμόσαμε, αλλά ένα από τα πλεονεκτήματα του Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση είναι η ευελιξία μεταφορά κοντιλίων από τη μία γραμμή του προπολογισμού σε άλλη εάν αλλάξουν οι συνθήκες. Π.χ. αν ε, τα λόγα άτομα αλλάξουν άποψη και θέλουν τελικά να ανοίξουν μια επιχείρηση, αυτή η ευελιξία μας βοηθάει στην εφαρμογή όμως κάποια από τα πλεονεκτήματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ήταν η διαδικασία η οποία παίρνει πάρα πολύ χρόνο, η διαδικασία έγκρισης των αιτήσεων. Βεβαίω δεν υπάρχει κάποια συνταγή για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα όπως επίσης και το θέμα της εθνικής συνεισφοράς και αν ένα κάποιο κράτος μέλος δεν έχει να συνεισφέρει τα κονδύλια εξ αρχής ε, τελικά δεν θα κάνει αίτηση γιατί θα περιμένει πάρα πολύ χρόνο ο κόσμος για τα κονδύλια του. Οπότε θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα από το να περιμένουμε στήριξη από το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση, γιατί για τον κόσμο δεν έχει διαφορά από πού θα πάρει τα λεφτά. Δεν κάνει διάκριση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση. Έλεγα λοιπόν πως είναι ευκολότερο και απλώς να χρησιμοποιήσουμε το ΕΚΤ βεβαίως σε καιρούς οικονομικής κρίσης όταν μια χώρα κάνει τον προϋπολογισμό της αναζητά ευκαιρίες να χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές και το ΕΚ είναι μια κάποια στήριξη και το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Αυτή είναι η απόψή μας γι' αυτό. Συνοψίζοντας λοιπόν θα ήθελα να κάνω κάποιες προτάσεις και να επισημάνω πως ε, η Λιθουανία έχει ακόμα μια επιφύλαξη εξέτασης για τον νέο πανίσμα γιατί η επέκταση του πεδίου εφαρμογή και η εμπλοκή νέων ομάδων του πληθυσμού είναι κάτι το οποίο ακόμα ε, συζητάμε. Κάποιοι λένε πως ε, είναι καλό να συμπεριληφθούν οι αγρότες, αλλά αν το δούμε ευρύτερα, μπορούμε να ρωτούμε είναι θετικό αυτό σε τι διαφέρουν οι αγρότες από τους άλλους. Μήπως έχουμε διακριτική μεταχείριση ε, κατά των υπολείπων απολυμένων. Τώρα δεν θα μπω πολλές λεπτομέρειες ε, όσον αφορά τις προτάσεις που έχει κάνει η Λιθουανία αλλά νομίζω πως ε, το 50% απασχολησιμότητας που αναφέρεται ε, δεν είναι πολύ καλή πρόταση. Επίσης έχουμε και μία ερώτηση για το ποσοστό συγχρηματοδότησης ε, 65% γιατί η Κομισιόν θα κρίνει το εάν θα είναι 65% ή λιγότερο οπότε δεν μπορούμε να πούμε πως είμαστε υπέρ όλων των αλλαγών ε, στον κανονισμό. Οπότε Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μας και είμαι στην διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Περνάμε στο τελευταίο μας ε, προσκεκλημένο, τον κύριο Βάρκο Αγκούσνα, πρόεδρο της ομάδα των ε, Ευρωπαϊκών ε, Ταμείων στο Υπουργείο Ελευθερίας και Κοινωνικών Υποδέσεων στη Γερμανία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. 15 ε, χρόνια παρακολουθούσα την ε, Επιτροπή ω σύνδεσμος ε, του Υπουργείου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα είμαι εδώ πέρα από τη νέα μου ιδιότητα και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι έχω 10 λεπτά χρόνο γιατί είναι πάρα πολύ σπάνιο αυτό. Συνήθως οι εισηγητές έχουν 3 λεπτά να μιλήσουν. Θα ήθελα τώρα να αναφέρω τις ε, εμπειρίες της ε, εφαρμογής ε, του Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση στη Γερμανία και συγκεκριμένα τι ποσοστά έχουμε επιτύχει στην επανενσωμάτωση. Εδώ πέρα βλέπουμε τα έργα τα οποία ξεκινήσαμε στο πλαίσιο του Ταμείου. Βλέπετε BNQ, Nokia, Carman, Heidelberger Druck, για να αναφέρω κάποιες. Αυτή τη στιγμή έχουμε υποβάλει πέντε αιτήσει, έχουμε 6.700 εργαζόμενους που έχουν επηρεαστεί. Από αυτούς μαζί με τα μέσα του Ταμείου ε, βρήκαμε εργασία σε 3.900, μιλάμε δηλαδή για ένα ποσοστό επανένταξη στην αγορά εργασίας 58%. έχουμε μία διακύμανση από 30 έως 80 της 100 ε, και αυτό ε, βεβαίως ε, εξαρτάται από την συγκυρία και τα προσόντα δεν σημαίνει πως όλοι θα επενταχθούν αυτομάτως στην αγορά εργασίας, εξαρτάται από το επίπεδο εκπαίδευσης. Η εμπειρία μας είναι πως αυτοί οι οποίοι έχουν πιο πολλά προσόντα έχουν ε, βεβαίως και μεγαλύτερη ετοιμότητα να εκπαιδευτούν περισσότερο ε, και άρα στο πλαίσιο του ταμείου αυτού έχουμε διαφορετικά μέσα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να στοχεύσουμε και τις διάφορες ομάδες καλύτερα. Συνολικά μπορούμε να πούμε πως το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης ε, νομίζω πως είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στη Γερμανία Τώρα τι, πώς χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα τα μέτρα αυτά. Ξέρετε πως ε, από πλευράς ε, μέσων ε, αγοράς εργασίας που έχουμε στη Γερμανία είναι θα έλεγα το κερασάκι στην τούρτα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Γιατί, γιατί έχουμε μια ολόκληρη σειρά ε, μέσων αντίδραση σε μεγάλες απολύσει ή κύματα απολύσεων. Αναφέρω δύο από αυτά. Το ένα είναι το ότι συμμετέχουν ε, οι εταίροι της επιχείρησης στον προγραμματισμό και των απολύσεων, κάτι το οποίο είναι βεβαίως στοιχειώδες. Μετά υπάρχει ε, μία σειρά μέσων κονδυλίων ουσιαστικά θα αναφέρω μόνο το εθνικό κοινωνικό τέτοιο σχέδιο το οποίο έχουμε και βεβαίως έχουμε διάφορα υποστηρικτικά μέτρα. Δηλαδή, γι' αυτό μίλησα για το κερασάκι στην τούρτα, γιατί μας προσφέρει την δυνατότητα να ενισχύσουμε παροχές που ήδη έχουμε Υπάρχει επίσης μια χρονική επέκταση της στήριξης των διαφόρων επιδομάτων και βεβαίως ε, στο πλαίσιο του Ταμείου για την έχουμε την δυνατότητα να αναπτύξουμε δοκιμασμένες ε, πρακτικές ή να αναπτύξουμε νέες ε, προσεγγίσεις. Οπότε έχουμε και συμβουλές και επανεκπαίδευση για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ακολουθήσουν νέες σταδιοδρομίες. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που άλλαξαν τελείως σταδιοδρομία, έκαναν ακολούθησαν ένα τελείω διαφορετικό κλάδο, άλλοι αποφάσισαν να ξαναμπούν στην εκπαίδευση, να σπουδάσουν, οπότε το εύρος ε, είναι πάρα πολύ μεγάλο των επιλογών, άλλοι έκαναν μία περαιτέρω μετεκπαίδευση στον ε, τομέα τους, οπότε μπορεί το Ταμείο να χρησιμοποιηθεί υποστηρικτικά για να επεκτείνουμε το χρόνο εφαρμογής αυτών των μέτρων. Οπότε, όπως είπα, μπορεί να μας βοηθήσει το Ταμείο για την παγκοσμιοποίηση, ειδικά για άτομα τα οποία είναι πιο ηλικιωμένα, έχουν λιγότερα προσόντα και αυτό μας έδειξε η μεσοπρόθεσμη αυτή αξιολόγηση, την εφαρμογή στα κράτη-μέλη το καταλάβατε βεβαίως διαφέρει πάρα πολύ και συνολικά θα έλεγα πως ε, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε ένα επίπεδο επανένταξης γύρω στο 11% και θα έπρεπε βεβαίως να αυξηθεί το 11% είναι απογοητευτικό αλλά το ακούσατε αποφασιστικής σημασίας είναι ε, το τι γίνεται και στην εθνική αγορά εργασίας και βεβαίως αυτή η αποχώρα από κράτος μέλος κράτος μέλος διαφέρει και διαφορετική επίσης είναι η εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη στη Γερμανία είναι βασικό στοιχείο των ε, μέτρων μας και στο πλαίσιο του Ταμείου για την παγκοσμιοποίηση δηλαδή τα κράτη-μέλη ε, αν θέλουν να αναπτύξουν περαιτέρω το Ταμείο αυτό πρέπει να σκεφτούν και την εθνική τους πολιτική εργασίας για να μπορέσουν να ε, εντάξουν καλύτερα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την παγκοσμιοποίηση. Ένα σημείο κριτικής είναι η εμπειρία που είχαμε πως ε, κατ' ουσίαν το Ταμείο αυτό το έχουμε σκεφτεί ως ένα μέσο παρέμβασης στην κρίση. Και βεβαίως για εμάς ε, μεγάλη σημασία έχει η διαδικασία ε, η, η αίτηση η οποία κρατάει 9 με 11 μήνες. Είναι πάρα πολύ μακροσκελής γιατί σας το λέω ανοιχτά, δεν θα υπέβαλε τη η Γερμανία αν δεν είχαμε, όπως σας είπα, τα μέσα τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αυτός ο χρόνος και πρέπει να δούμε πώς θα απλοποιηθεί αυτή η διαδικασία και να μειωθεί αυτός ο χρόνος. Όπως είπα, για τη Γερμανία ανέφερα πως είναι ένα συμπληρωματικό μέτρο δεν είναι κάτι το απολύτω απαραίτητο το ταμείο αυτό. Τώρα να έρθουμε για, την, ε, για τις, προτάσεις, τις Κομισιόν. Υπάρχει ένα λάθος εδώ πέρα στη σκέψη της Κομισιόν γιατί βλέπουμε πως ε, υπάρχει μόνο μία απορρόφηση 10 με 15% των διαθέσιμων κονδυλίων. Όταν έχουμε κάτι τέτοιο και βλέπουμε Πω δεν απορροφούνται τα κονδύλια. Πρέπει να σκεφτεί κανεί διαρθρωτικά ποια είναι τα προβλήματα, γιατί δεν απορροφούνται αυτά τα κονδύλια. Κατά την άποψή μα, λοιπόν η Κομισιόν κάνει, ε, ακολουθεί μια λανθασμένη πορεία, δηλαδή πηγαίνει και προσπαθεί να επεκτείνει το εύρος των ε, ομάδων που εποφελούνται από ε, το Ταμείο Προσαρμογής. Ε, εάν δούμε δε τους ε, γεωργούς που λαμβάνουν λεφτά από 5-6 διαφορετικές πηγές, νομίζω πως δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε περαιτέρω με αυτούς. Νομίζω λοιπόν πως θα έχουμε φτάσει σε σημείο παράλογο. Δηλαδή έχουμε φάλει μέσα και τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους και τι θα γίνει μετά. Ε, το αρχι η αρχική ομάδα στόχος ε, θα έχει απομείνει με το 1 έκτο του Ταμείου και δεν θα το αναγνωρίζουμε σε σχέση με τον αρχικό του σχεδιασμό. Μπορεί βεβαίως κανείς να πει το επιχείρημα πως ε, στο πλαίσιο των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου επιβαρύνεται πάρα πολύ η γεωργία, αλλά κοιτάξτε, τότε μπορούμε να το πούμε και να το ορίσουμε ως ένα μέσο της ε, γεωργίας. Δεν είναι πλέον μέσο της γενικότερης αγοράς ε, εργασίας. Το έχουμε αλλάξει τελείως. Επίσης, όσον αφορά την έννοια της κρίσης, η οποία επιχειρείται να εισαχθεί, είναι τόσο ασαφής έτσι ώστε το εύρος εφαρμογής ε, του Ταμείου διευρύνεται πάρα πολύ και πλέον δεν μιλάμε για κάτι το συγκεκριμένο. Γι' αυτό η Γερμανία ειδικά στο Συμβούλιο λέει πως το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης δεν το θέλουμε να έχει αυτή τη μορφή. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ένα σημείο δεν θίξατε. Που αφορά την παράταση του μηχανισμού αντιμετώπισης της κρίσης ε, στο πλαίσιο του παλιού συστήματος, διότι η Γήτρια έδειξε το ζήτημα αυτό. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει ήδη εκφραστεί υπέρ. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να επανέλθετε. Αλλά θα σας δώσω το λόγο φυσικά για να απαντήσετε στο σύνολο των ερωτήσεων. Ποιος επιθυμεί να θέσει ερωτήσεις. Μπάουερ, Μπλεκεβίτσι, Νταρντέν. Monsieur Sarkas, Madame Pérez et la rapportrice. Voilà, alors on va commencer. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την κυρία Μπάμπα. Αυτές οι παρουσιάσεις ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Έχω τρεις ε, σύντομες ερωτήσεις ε, σχετικά με τη χρηματοδότηση. Ποιες είναι οι εμπειρίες που έχετε με τη χρηματοδότηση. Ποιες είναι οι πηγές που χρησιμοποιείτε για κάτι τέτοιο. Το δεύτερο ερώτημα αφορά την γεωργία. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε πόσα θα είναι τα χρήματα που θα προωθηθούν στην Γεωργία. Δεν μου φαίνεται ότι είναι σωστό από αυτό το ταμείο να χρηματοδοτήσουν και τους ε, καλλιεργητές και τους γεωργούς. Τρίτη ερώτηση. Στην τελευταία παρουσίαση ακούσαμε ότι θα πρέπει να ε, εναρμονιστεί το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης και το Κοινωνικό Ταμείο. Πού βλέπετε να υπάρχει δυνατότητα τέτοια είδου εναρμόνισης. Κύριε Λικεβιτσούρη, κύριο Νταρδέν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Ήταν πολύ χρήσιμο να ακούσουμε τις εμπειρίες των πρωτομελών από την χρησιμοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν μιλάμε και για τις μελλοντικέ προοπτικές. Θα ήθελα τώρα να τονίσω πως το Ταμείο Προσαρμογής, την παγκοσμιοποίηση, χρησιμοποίησε το 15% των κονδυλίων και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο δείχνει ότι εάν ότι κάποιοι κανόνε ε, θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότερη απορρόφηση. Και τα κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν ε, μεν σε κάποιου κλάδου αποτελεσματικά τα κονδύλια αυτά. Και έχω όμω κάποιε ερωτήσει. Όταν αποφασίσουμε πω το Ταμείο Προσαρμογή χρειαζόταν, δεν κρίνεται ότι το κατόφλι των 500 εργαζομένων δεν είναι μια κατάλληλη παράμετρος ε, ειδικά όταν βλέπουμε μεγαλύτερα κράτη-μέλη, χρειάζεται να βρούμε τρόπο να βοηθήσουμε αυτούς τα άτομα που χάνουν την εργασία τους, που απολύονται. Βλέπουμε ότι το Ταμείο Προσαρμογής έχει ικανούς πόρους, εκτός εάν ο τομέας Γεωργίας πάρει το μεγαλύτερο τμήμα αυτών, ίσως ε, θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το ποσοστό του 65% στο 75% και η τρίτη μου ερώτηση αφορά στο ότι υπάρχουν νέες ε, απαιτήσει ε, σχετικά με το 50% των προσώπων που βρίσκουν επανεπασχόληση μετά από 12 μήνες. Αλλά τι είδους απασχόληση είναι αυτή, είναι μόνιμη εργασία, είναι ποσορινή Γιατί να μην συμπεριλάβουμε την περίοδο της κατάρτισης, της εκπαίδευσης αυτή την χρονική περίοδο των 12 μηνών και μια ακόμα ερώτηση που αφορά στη Γεωργία γιατί θέλουμε να συμπεριλάβουμε την μάλλον να αποφασίσουμε να συμπεριλάβουμε τη γεωργία τότε θα πρέπει οι κανόνες να είναι αυτοί όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά Εάν πολλοί εργαζόμενοι χάσουν την δουλειά τους σε αυτόν τον κλάδο, θα μπορούσαν ε, να επιλεγούν για να χρησιμοποιηθεί το κονδύλι για αυτούς. Αλλά τότε δεν εμπίπτει στη δική μας αρμοδιότητα το ζήτημα, δική μας επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες ε, για τις μαρτυρίες τους. Ε, τίνω να πω ότι χαίρομαι με τις μαρτυρίες αυτές ε, που ενδυναμώνουν την άποψή μας ε, και την αναγκαιότητα του Ταμείου. Ακούσαμε τα παραδείγματα που αφορούσαν πολλούς εργαζόμενους. Φυσικά δεν επέτρεψε το πρόγραμμα σε όλους να βρούνε εργασία, εργασία. Με βάση τα όσα άκουσα λοιπόν, είναι σαφές πως το κριτήριο της κρίσης ε, διατηρεί τη σημασία του, διότι ε, όλοι οι φάκελοι είναι φάκελοι που αφορούν ε, στην κρίση. Άκουσα επίσης με χαρά την εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων. Είναι κάτι που μας απασχόλησε Γι' αυτό και ανηφέραμε ότι θα πρέπει να τονίσουμε περαιτέρω το ζήτημα στο νέο κανονισμό, να υπάρξει μια, ένα σημαντικό ύψος συγχρηματοδότησης. Έχω δε την εντύπωση πως ε, συμφωνούμε ώστε η επέκταση στο γεωργικό τομέα δεν είναι σκόπιμο. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε το ζήτημα εδώ στο κοινοβούλιο μας Να διευκρινίσουμε επίσης και τις αρμοδιότητες ε, των ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών και να παραμείνει ένα θέμα που αφορά στην απασχόληση και όχι το σύνολο, το στην ε, επεκταθεί δηλαδή στη γεωργία και κάτι ακόμα να μειωθεί η διάρκεια διάρκεια εξέταση και επεξεργασία των φακέλων ε, να μην περνάει πολύς χρόνος ανάμεσα στην απόλυση και την παρέμβαση της ε, Ένωσης ε, και του Ταμείου. Η ερώτησή μου είναι εξή. Τι προτάσεις έχετε προκειμένου να μειωθεί αυτή η προθεσμία και άλλη μια ερώτησούλα αφορά την παρέμβαση του Γερμανού εμπειρογνώμονα Συμφωνώ με την παρέμβασή του, αλλά ξεπλάγει από το συμπέρασμα ότι με αυτή τη μορφή δεν θέλουμε πλέον το Ταμείο. Υπό ποια μορφή το επιθυμείτε, διότι μπορεί να μην είναι τέλειο, άρα μπορούμε να το βελτιώσουμε, αλλά να το καταργήσουμε θεωρώ πως θα ήταν σφάλμα. Θα ήθελα λοιπόν μια διευκρίνηση στο σημείο αυτό. Σέρκας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους τρεις ε, εμπειρογνώμονες, ε, διότι αναφίβολα θα μας βοηθήσουν πολύ στις εργασίες μας της προσεχής εβδομάδας. Να κάνω δύο ερωτήσεις, τον Γερμανό και τον Ισπανό εμπειρογνώμονα. Και ως εκ τούτου να διευκνήσουν δύο ζητήματα που θεωρώ ενδιαφέροντα. Στη Γερμανία ακούσαμε ότι η ε, ε, γίνεται, εφαρμόζεται με τρόπο συλλογματικό παράλληλα με άλλες εθνικές πολιτικές στον τομέα της αναδιάρθρωσης. Αυτό είναι ένα θέμα κλειδί το οποίο κατέδειξε την αποτελεσματικότητα. Θα θέλω να γνωρίζω πώς ε, χρησιμοποιούν το Ταμείο και πώς συνδέεται με τις εθνικές πολιτικές τώρα στον Ισπανό συνάδελφο ε, εμπειρογνώμου, να τον ευχαριστήσω για το ότι μας μίλησε για την φοβερή προσπάθεια που καταβάλει για την διάσωση θέσεων απασχόλησης ε, στην χώρα μου που πλήττεται από την κρίση. Να μας πει κάτι για τη Γεωργία. Εγώ δεν ε, έχω αντίρρηση να δοθεί ένα ποσοστό και στον τομέα της γεωργίας. Ε, η, γεωργία είναι, η Ισπανία είναι αυτή η οποία παίρνει τα δεύτερα σημαντικότερα ποσά από το, στον τομέα της γεωργίας, ε, ο οποίος ε, πλήττεται σημαντικά με το άνοιγμα των αγορών, την κατάργηση των δασμών κλπ. Τι θα συμβεί στην Ισπανία, κύριε Τοτουέρο, εάν αυτά τα χρήματα χορηγηθούν και στο Υπουργείο Γεωργία στην πράξη, τι θα συμβεί. Θα ήθελα λοιπόν να διακινδυνεύσετε κάποιος και να μας πείτε τι θα συμβεί με το Ταμείο, εάν γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πέραν του ε, παράτασης του μηχανισμού. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο-τρία σημεία. Μας είπατε, εννέα μήνες είναι υπερβολικά μακρύ χρονικό διάστημα. Τι θα προτιμούσατε λοιπόν ως προθεσμία. Και συμφωνούν οι άλλοι δύο εμπεροχνόμενες με τη μείωση της προθεσμίας αυτής. Και όσον αφορά την καθυστέρηση της εφαρμογής, γιατί υπάρχει περίπτωση παρακολούθησης, μετά υπάρχει η προθεσμία για την κινητοποίηση του Ταμείου και για την κινητοποίηση αυτή, κυρία ναι. μας είπε ότι το ε, κοινωνικό ταμείο ήταν καλύτερα. Γιατί είναι καλύτερο να αφορά τις προθεσμίες. Κατόπιν. Έχω μία σειρά παρατηρήσεων και για τους τρεις υπερογνώμονες. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να οριστεί ένα όριο ηλικίας για τους δικαιούχους ε, του Ταμείου, γιατί ο στόχος του Ταμείου είναι η επανακινητοποίηση των ε, εργαζομένων. Δηλαδή να έχουν μια μεταβατική περίοδο για το, ε, ε, να απασχοληθεί τους. Γιατί εγώ είδα ότι υπήρχαν ηλικιωμένοι εργαζόμενοι σχεδόν σε ηλικία της και τους μαθαίνανε πώς να σκαλίσουν στον κήπο ή να ζουν μια υγιεινή ζωή. Ε, δεν είναι λογικό αυτό, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Κατόπιν, στα δύο κριτήρια κινητοποίησης ε, του Ταμείου υπάρχει το θέμα κατά πόσο πλήττεται μια περιοχή ή μια συγκεκριμένη ε, επιχείρηση και ξέρουμε ότι στη Γερμανία με οποίο υπάρχει πολλές φορές η εντύπωση ότι στην πραγματικότητα σε αυτού του τύπου την ε, κινητοποίηση του ταμείου Μια συγκεκριμένη δηλαδή επιχείρησης κατά βάση το ταμείο αυτό χρησιμοποιείται για την μεταφορά τη γεωγραφική ολόκληρης μιας πολυεθνικής εταιρείας δεν ξέρω, μήπως θα πρέπει να οριστούν κάποιοι άλλοι όροι. Καταλαβαίνετε δηλαδή την σχέμα, αν πρόκειται για μια πολυεθνική εταιρεία θα πρέπει τα προγράμματα του, να, του ΦΕΜ να εφαρμοστούν του, και να ζητήσουμε όμως από την πολυεθνική να πληρώσει ε, εκτός από τα μέσα συνοδείας των εργαζομένων και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προβλέπετε. Εσείς ε, πώς τη βλέπετε αυτή την πρόταση. Δεύτερη σειρά ερωτήσεων. Αφορά ακριβώς τις πληροφορίες που μπορεί να δοθούν για τη λειτουργία του Ταμείου σχετικά με το Κοινωνικό Ταμείο. Γνωρίζοντας ότι όπως κατάλαβα, έχω την εντύπωση ότι στο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης προβλέπονται συνοδευτικά μέτρα για άτομα που είναι πολύ πιο, πιο συγκεκριμένα τα μέσα αυτά, πιο συγκεκριμένα για το κάθε άτομο που ωφελείται. Το βλέπετε αυτό επί τόπου πραγματικά έτσι. Τελευταία ερώτηση. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο διατήρηση τακτικό για τη χρησιμοποίηση αυτών των προβλέψεων της νομοθεσίας για να μπορέσουν καλύτερα να οριστούν τα διάφορα μέτρα που υπάρχουν για τη συνοδεία των εργαζομένων και την κινητοποίηση της μικρό χρηματοδότησης που προβλέπεται στα ευρωπαϊκά προγράμματα για να βοηθηθούν ακριβώς εκείνοι οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν στην ε, ίδρυση μιας επιχειρήσης ή οτιδήποτε άλλο. Παρακαλώ. Thank you, Madam, Κύριε Συγκήτρια, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους τρεις εμπειρογνώμονες. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είπατε. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα στον ε, συνάδελφο από την Ισπανία, τον Κάρλος. Με ενδιαφέρον είδα πως στην Ισπανία πέντε από τις παρεμβάσεις ε, οφειλόταν στην ε, παγκοσμιοποίηση και 13 στην κρίση και στη Λιθουανία 41. Οπότε βλέπουμε την ανάγκη να συνεχιστεί η παρέκκληση της κρίσης. Δεν ξέρω ποια ήταν τα νούμερα στη Γερμανία. Θα μπορούσε ίσως ο κύριος να μας διαφωτίσει. Και πάλι προς τον Ισπανό συναλφό είπατε πως θέλετε θέλατε να συνεχιστεί το κεφάλαιο της κρίσης και μιλήσετε για 65% χρηματοδότηση που χρειάζεται αυτό θα είναι διαθέσιμο με τη νέα πρόταση αν έχει ε, μια περιοχή επιλέξιμη ένα κράτος μέλος. Ε, νομίζω αυτό θα γίνει στην Ισπανία. Επίσης μιλήσατε για αλλαγή του αριθμού των εργαζομένων που καλύπτονται και αναρωτιέμαι θεωρείτε πως το άρθρο 4.2 δεν είναι αρκετά ευέλικτο γιατί λέει σε μικρές αγοράς εργασίες, εξαιρετικές συνθήκες κτλ μπορεί να υπάρξει παρέκκληση από τον αριθμό των 500. Εκεί όπου υπάρχει σοβαρή, σοβαρός αντίκτυπος στην ε, αγορά εργασίας της τοπικής οικονομίας. Είναι αρκετά ευέλικτο ή θέλετε κάτι πιο ευέλικτο. Και δύο ακόμα ερωτήσεις. Ξεκινήσατε τις παρεμβάσεις μόλις κάνατε την έτσι ή περιμένατε να λάβετε τα χρήματα. Και ποιο μέρος των χρημάτων που χρησιμοποιήσατε στην συνάδελφο από τη Λιθουανία. Είπατε πως ε, τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά σε διαφορετικές συνθήκες. Ποια ήταν τα βασικά ζητήματα που επηρέασαν ε, διαφορετικά αποτελέσματα. Δεύτερον, θέλω να ξέρω, ξεκινήσατε αμέσως τις ε, πρωτοβουλίες. Γιατί αναφέρατε πως τα κονδύλια αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα. Χρησιμοποίησατε ένα συνδυασμό ταμείων για να βοηθήσετε τους απολυμμένους εργαζόμενους. Και υποθέτω πως το ποσοστό συγχρηματοδότησης, θα μας πείτε ποιο είναι, αλλά υποθέτω πως είναι μεγαλύτερο του κοινωνικού ταμείου από το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Έκανε αυτό διαφορά. Επίσης μιλήσατε για την επέκταση του πεδίου εφαρμογή και πως είναι συζητήσιμο το εάν πρέπει να συμπεριληφθούν οι ευρώτες. Και έχω μια ερώτηση και για τους τρεις σας. Τέλος, το τη Γερμανία, με χαρά άκουσα ήταν υποδειγματικά τα αποτελέσματα στη Γερμανία. Αυτό α, παντού ακούω, αλλά χαίρομαι που το λέτε κι εσείς. Μιλήσατε για τον χρόνο, βεβαίω την έγκαιρη παρέμβαση, αλλά λέτε πως η Κομισιόν έχει, λάβει, έχει κάνει λάθος προσέγγιση με την επέκταση και στους αγρότες. Έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, θεωρείτε πως πρέπει να συμπεριληφθούν οι αγρότες. Δεύτερον, εάν συμπεριληφθούν να είναι με, στην ίδια βάση με τους άλλους εργαζόμενους ή σε διαφορετική βάση. Και εάν είναι σε διαφορετική βάση ε, θα πρέπει η Κομισιόν να αποφασίσει στα κριτήρια αυτά με πράξη κατά εξουσιοδότηση. Και τέλος, αναφερθήκατε ήδη στα ποσά, αλλά αν θέλετε να το ξανακάνετε. Τέλος, ε, ο κ. από τη Γερμανία μίλησε για την κρίση και πως στο νέο κανονισμό ε, ήταν πολύ ευρύς ο ορισμός θα ήθελα να ξέρω πώς ε, θεωρείτε, πώς μπορεί να το συμμαζέψουμε αυτό εδώ πέρα. Έχοντας μιλήσει με την Κομισιόν για το άρθρο 2β, μιλάνε για εργαζόμενους που απολύονται λόγω σοβαρών ε, προβλημάτων στην τοπική εθνική οικονομία λόγω κρίσης η οποία δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Π.χ. πλημμύρες σε μια περιοχή μπορούν να καταστρέψουν μια επιχείρηση, ένα σύννεφο τέφρας μπορεί να κλείσει μια αεροπορική εταιρεία. Ε, πώς πρέπει κατά την άποψή να αλλάξει ο ορισμός ε, της κρίσης που έχουμε εδώ και ποιο θα ήταν το πλεονέκτημα. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι οι τρεις εμπειρογνώμενες σημείωσαν όλες τις ερωτήσεις και σε πέντε λεπτά θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις αυτές. Πρώτον, να ακολουθήσουμε την ίδια σειρά. Κύριε e, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ όλες αυτές ε, ερωτήσεις που βεβλήθησαν. Θα συγκεντρώσω την προσοχή μου στις κύριες ε, ερωτήσεις, δεν θα μπορέσω φαντάζομαι να απαντήσω σε όλες αυτή τη στιγμή. Η χρηματοδότηση 65% είναι καλύτερη από το 50%. Ναι. Και 85% βέβαια ε, για το από το κοινωνικό ταμείο είναι ακόμα καλύτερο. Για ε, τη αυτά τα στοιχεία. Όπως είπε ο βουλευτής ε, σωστά, αυτή τη στιγμή η Λουθανία χρηματοδοτείται από την, το κοινωνικό ταμείο με συγχρηματοδότηση τάξη του 85%. Πολύ καλό αυτό και η Λιθουανία χρησιμοποιήσει αμέσως τα μέσα παρέμβασης κατά διάρκεια της ε, υποβολής ε, των αιτήσεων γιατί χρησιμοποίησαμε ακριβώς ε, τα χρήματα από το Ταμείο Απασχόλησης από τον Εθνικό Προπολογισμό αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τα διάφορα σχέδια. Λοιπόν, θα ήθελα να σημειωθεί ότι προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε μια σειρά πηγών χρηματοδότησης από το Κοινωνικό Ταμείο, από το Ταμείο ε, Απασχόλησης. Τι θα μπορούσε να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση και πώς θα μπορούν να μειωθούν οι προθεσμίες. Εγώ ξέρω ότι στην Λουθανία ε, χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο για να αξιολογήσουμε τις ε, αιτήσει. τρει μήνες θα ήταν νομίζω θαυμάσιο, ιδανικό. Αν εγώ ήθελα να αποφασίσω και μόνο η αξιολόγηση των ε, προβλημάτων ε, παίρνει χρόνο. Όταν ε, εξετάζουμε βέβαια και αξιολογούμε το κάποιες επιχειρήσεις ενός τομέα μπορούμε να συμπεριλάβουμε και άλλες επιχειρήσεις. Ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε όχι μόνο μία επιχειρήση αλλά περισσότερες μία επιχειρήσεις του ιδίου τομέα χρησιμοποιώντα του πόρου του Ταμείου. Θα ήταν πολύ καλό αυτό, θα είχαμε μεγαλύτερη ευελιξία. Ο γερμανός συνάδελφος είπε ότι δεν συγκεντρώνουμε προσοχή μα στην επίλυση των προβλημάτων, δεν είμαστε αρκετά συγκεκριμένοι. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στο κεφάλαιο 4 και το κατόφλι των 500 εργαζομένων. Ο σημερινός κανονισμός ο κοινωνικός κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα να υποβληθεί αίτηση με χαμηλότερο ρυθμό εργαζομένων. Αλλά όταν μιλάμε για απολύσεις, 500 για τη Λιθουανία, όπως λέγεται στο οργανισμό, πρέπει να τηρηθεί. Γιατί αυτό το κατόφλι όμως είναι τεράστιο για τη Λιθουανία. Γιατί μόνο 1,2% όλων των επιχειρήσεων της χώρας απασχολούν πάνω από 500 εργαζόμενους. Είναι τεράστιο λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Αναφερόμενοι τώρα στη Γεωργία, ίσως δεν σας πω τίποτα καινούριο, γιατί το ανέφερα εισαγωγικά, το γιατί χάνουν τη δουλειά τους οι αγρότες για την κρίση, λόγω επικείμενης κρίσης είναι όλοι καταγραμμένοι στα ταμεία εργασίας και θα θεωρηθούν ότι έχουν απολυθεί και θα πάρουν όλα τα επιδόματα της κοινωνικής ασφάλειας που προβλέπει ο νόμος. Γι' αυτό η Λουθιανία δεν σημαίνει ότι είναι δυνατόν να υπάρχει μια ξεχωριστή κατηγορία για τους ε, περιτούς αν θέλετε απολυμμένους Γιώργους. Ελπίζω να ε, απάντησα στις ερωτήσεις. Αν ξέχασα κάτι μου το επιθυμίστε παρακαλώ. Merci. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάρλος Τορτουέρο έχει το λόγο. Sí, eh, Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στο μεγαλύτερο αριθμό ερωτήσεων που τέθησαν. Υπήρξε αναφορά. Παρακαλεί τον μιλητή να μιλά λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, να τον ακούμε. Τώρα, για τις πηγές χρηματοδότησης. Αυτές χορηγούνται από τους προπολογισμού των αυτόνομων κοινοτήτων. Η συγχρηματοδότηση γίνεται μετά από σύμβαση που υπογράφεται από το Ταμείο και τους υπευθύνους πολιτικών απασχόλησης σε αυτόνομες κοινότητες σε μερικές περιπτώσεις και σε άλλες από άλλους εμπλεκόμενους. Υπάρχει λοιπόν μια συνεισφορά περιφερειακού χαρακτήρα. Η χρηματοδότηση γίνεται από την περιφέρεια και όχι ο κεντρικός προϋπολογισμός του κράτους σου. Σχετικά τώρα με τα γενικότερα ζητήματα τα οποία ετέθησαν. Πώς ε, ε υπάρχει, ποια είναι η συμπληματικότητα που υπάρχει. Κατά άποψή μας, ε, ε, δύο αυτοί, τα δύο αυτά ταμεία, δηλαδή το Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Προσαρμογής, το Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα ταμείο διαρθρωτικό το οποίο αφορά στο σύνολο των ε, πολιτών ε, και, και επιθυμεί να βελτιώσει τις, ε, τα προσόντα, την κατάρτιση. Έχει το, λοιπόν το Κοινωνικό Ταμείο μια στρατηγική σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε πολυετή βάση και ε, οργανώνει τους στόχους τους, τους στόχους του ανάλογα κατά πόσον έχουν εκπληρωθεί ή όχι. Τώρα, ενώ το Ταμείο προσαρμογής είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Ένα ταμείο δράσης, βραχυπρόθεσμης, άμεσης δράσης ε, και προσπαθεί να αποφύγει την διόγκωση ενός ε, προβλήματος ε, και λειτουργεί σε μηχανισμό όταν ένα σημαντικός αριθμός εργαζομένων χάνει την δουλειά του. Τα δύο λοιπόν ταμεία το, λειτουργούν συμπληρωματικά και ο καθένας, το καθένα στον κλάδο του. Η εμπειρία στην Ισπανία σχέση με την ε, περίοδο ορίμανσης ε, της ε, βοήθειας που χορηγεί το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης είναι μια περίοδος ιδιαίτερα μακρά προκειμένου να ληφθούν αυτά τα κονδύλια. Η περίοδος ορίμανσης λοιπόν και η περίοδος των εσωτερικών διαδικασιών που το χρόνο περνάει από την υποβολή των αιτήσεων, των προγραμμάτων, τις συζητήσει ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και των Κομισιών έχουν ως αποτέλεσμα τα προγράμματα αυτά να μην ε, εφαρμόζονται άμεσα όπως προτίθεται να το πράξει το Ταμείο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες δράσεις ε, που προκαταβάλλονται στις ε, στις ε, αυτονόμες ε, κοινότητες. Στην Ισπανία η κάθε κοινότητα έχει το δικό της ε, επιχειρησιακό πρόγραμμα. τους οποίους χρηματοδοτεί με τα δικά της κονδύλια. Πάντως η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής όταν φτάσουν, όταν καταβάλει τα κονδύλια τότε συμπληρώνει αυτήν την ε, δράση και την συγχρηματοδοτή. Όπως είπαμε λοιπόν, ε, η δράση είναι συμπληρωματική και Μιλώντας τώρα για το ποσοστό συγχρηματοδότησης ε, κατά την άποψή μας, η κατάσταση η σημερινή που μας οδηγεί στο 50% είναι κάτι το οποίο δεν, μάλλον κρίνουμε το οποίο δεν μπορούμε να αναλάβουμε. Θεωρούμε ότι είναι μια υπαναχώρηση, μια οπισθοδρόμηση. Ε, όταν ε, ένα ταμείο δεν ε, μπορεί να χορηγήσει τους χώρους πόρους, ειδικά σε περίπτωση κρίσης και νομίζουμε ότι η προσαρμογή αυτού των ε, ταμείων στο 65% και αυτό είναι λίγο. Είχαμε μιλήσει για 75%. Μια μεγαλύτερη λοιπόν οικονομική συνδρομή θα βελτιώσει τα αποτελέσματα. Τώρα σε ό,τι φορά τον αριθμό των ε, εργαζομένων. Είπαμε 500, αλλά θα μπορούσαμε να ορίσουμε 300 εργαζόμενους. Στην Ισπανία ο, ο παραγωγικός ιστός, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις, ε, για να φτάσουν ε, τις απολύσεις 300 ε, ατόμων η κάθε μια, θα χρειαζόταν μια μεγαλύτερη συνδρομή με μεγαλύτερη στήριξη από το Ταμείο. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να μειωθεί αυτό το ποσό των 500 ε, τώρα. Να πω τώρα προς τον ε, Αλεξάνδρου Θέρκας ε, ότι τον ευχαριστώ για την επίσκεψη που μας έκανε στην Ισπανία με την Ευσοπία του Ευρωπαϊκού Να το απαντήσω για το ζήτημα της Γεωργίας. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί στο Ταμείο Προσαρμογής Παγκοσμιοποίησης ε, περιλαμβάνεται η Γεωργία. Από αυτή την άποψη ε, θεωρούμε ότι βρίσκεται εκτός ε, τόπου. Η αφορτική πολιτική έχει τους πόρους, έχει την παράδοσή του, έχει τις δυνατότητες, έχει τις ειδικέ δράσεις και δεν καταλαβαίνουμε πώς θα πρέπει να αφιερώσουμε ένα σημαντικό κομμάτι του Ταμείου Προσαρμογής στον γεωργικό τομέα. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα περιόριζε τις δυνατότητες δράσης ε, του Ταμείου. Εντάξει, ας υπάρξει ένα ειδικό Ταμείο για τη Γεωργία. Και ίσως ε, να μην χαθούν με αυτόν τον τρόπο πόροι, μάλλον δεν θα χαθούν πόροι, από το Ταμείο Προσαρμογή που αφορά τους υπόλοιπους τομείς. Εμείς λοιπόν ε, δεν στηρίζουμε να συμπεριληφθεί και η Γεωργία στο Ταμείο Προσαρμογής Παγκοσμιοποίησης. Ε, Αγαπητέ φίλε, αν θέλετε μία πρόταση να μας πει το βασικό μήνυμα, μετά πρέπει να περάσουμε στον τελευταίο εμπειρογνωμούνα μας. Το Ταμείο Προσαρμογής είναι ένα ταμείο πάρα πολύ σημαντικό για να βοηθήσουμε τα άτομα που έχασαν την δουλειά τους σε περίπτωση μαζικών απολύσεων. Πολύ σημαντικό λοιπόν και θα πρέπει να διατηρηθεί διευκολύνοντας ε, τα μάλα, την χρησιμοποίησή του, τη διαχείρισή του και επιτυχάνοντας μια μεγαλύτερη συμμετοχή όλων ε, των εμπλεκομένων τόσο σε κοινό επίπεδο όσο και σε περιφερειακό αλλά και φυσικά των ενδιαφερομένων και τη στήριξη όλων των ε, με τη στήριξη όλων των θεσμών. Ευχαριστώ κύριε Σώσο. Στα γλίγορα. <clears throat> λόγω της δημοκρατικής εξέλιξης στην Ευρώπη δεν μου φαίνεται ότι είναι χρήσιμο. Δεν ξέρω ε, τι θα μπορούμε να κάνουμε για να διευκολύνουμε την ε, μετάβαση στην ε, σύνταξη. Αυτό δεν ταιριάζει νομίζω με την εικόνα που θέλουμε να δώσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο όμω. Προθεσμίες. Υποβολή αίτηση. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε έξι μήνες ρεαλιστικά. η μεταφορά της, ε, του τόπου εγκατάστασης, στον οποίο αναφερθήκατε σε σχέση με την Όκια, ε, από έξω αυτή η εικόνα δίνεται, στη Γερμανία όμως είναι διαφορετική εικόνα. Θα πρέπει καταρχήν οι κοινωνικοί εταίροι στο επίπεδο της επιχείρησης να συμφωνήσουν για ένα κοινωνικό ε, πρόγραμμα, δηλαδή ακόμα και τον αριθμό των απολύσεων κλπ. Και μετά εμπλέκεται το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Πολλές επιχειρήσεις που πλήττονται από τις απολύσεις τα βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά, αλλά εμείς δεν έχουμε άμεση επαφή με τις επιχειρήσεις. Ε, τους λέμε ότι εντάξει, έχετε μια κρίση, ενδιαφέρον είναι, ας συμφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι της επιχειρήσης όμως πάνω σε ένα κοινωνικό πρόγραμμα και θα δούμε μετά πώς μπορούμε εμείς με τους πόρους από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης το Ταμείο της Εθνικής Πολιτικής να συνοδεύσουν τα μέτρα που αποφασίζεται. Και το Υπουργείο Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι υπεύθυνο για την υποβολή των αιτήσεων στο Ταμείο Παγκοσμιοποίηση και την εφαρμογή των αποφάσεων. Έχουμε μια συνεργασία με την Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόληση, που εάν έχουν συνοενωθεί οι κοινωνικοί εταίροι για το κοινωνικό πρόγραμμα, δίνει τη δυνατότητα σε μια μεταβατική εταιρεία να επιβάλλει κάποια μεταβατικά μέτρα. Δεν είναι λοιπόν σωστό αυτή η ιδέα που υπάρχει στην κοινή γνώμη ότι οι επιχείρησεις ε, μας έρχονται και μας λένε και προσπαθούν να δουν ποιου πόρους θα μπορούσαν να πάρουν και πώς με τη βοήθεια των πόρων αυτών θα μπορούσαν να απολύσουν περισσότερους. Ε, δεν θέλουμε να ευκολούν ζωή έτσι και γι' αυτό ακολουθούμε τη μέθοδο που σας αναφέρω εδώ και 7 χρόνια. Τι μπορούμε να μάθουμε από τη σχέση Ταμείου Παγκοσμιοποίησης και Κοινωνικού Ταμείου. αυτό που μπορούμε να μάθουμε από το Κοινωνικό Ταμείο σε σχέση και με τον νέο οικονομισμό είναι μεγαλύτερη συγκέντρωση και ακρίβεια της χρήσης των μέσων. Δηλαδή ακριβώς και το συγκεκριμένο ερώτημα ποια είναι η προστιθέμενη αξία που μας δίνει αυτό το μέσο. Με δύο λόγια δηλαδή, εμείς όσον αφορά το νέο κανονισμό του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης να διατηρηθεί ο προσανατολισμός που έχει για την απασχόληση. Και ακριβώς το Κοινωνικό Ταμείο κάνουμε το αντίθετο αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε δηλαδή να συγκεντρώσουμε τα διάφορα μέσα και να προσανατολιστούμε καλύτερα σε συγκεκριμένους ε, ομάδες του πληθυσμού στόχους. Και δεν θα πρέπει νομίζω να στραφεί το κοινωνικό ταμείο προς την εξυγχρονισμό και το ταμείο που χρησιμοποιήσει να πάει προς τα πίσω. Τώρα, χρηματοδότηση, συγχρηματοδότηση στη Γερμανία γίνεται μέσω των ε, χρημάτων ε, μεταφοράς για περιορισμένε ώρε εργασία. Εμεί δεν έχουμε συγκεκριμένου πόρου για τη διάθεση αυτό και στη διαδικασία που έχει προαναφερθεί μπορούμε πολλά μέτρα και μέτρα που αφορούν ομάδες και μετεκπαίδευση ολόκληρων ομάδων και συμφωνία με το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση. Κατά πόσο θα πρέπει να το διαγράψουμε το ταμείο αυτό, ένα θέμα που έθιξα προηγουμένω. Η θέση τη Γερμανία, αν κοιτάξει κανένα και την ιστορική αναδρομή, θα βλέπετε ότι το 2006-2007 η Γερμανία ήταν ήδη τότε κατά του ταμείου. Και όπως έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή, στο Συμβούλιο η Γερμανία, μπορώ να σας το πω ξεκάθαρα, θα καταψηφίσει και στη νέα μορφή, η λειτουργικά τροποποιημένη μορφή. Αυτό είναι που πρέπει να σας πω αυτή τη στιγμή για να σας παρουσιάσω τη γερμανική θέση σχετικά. Euh, Ευχαριστώ. Σας είχαμε ζητήσει αν αποδείξετε ότι στην Γερμανία χρησιμοποιείται πιο σωστά και αποτελεσματικά το Ταμείο. Νομίζω ότι η γερμανική εμπειρία θα μας κάνει να βγάλουμε κατάλληλα συμπεράσματα σχετικά με τα αλλαγές του νέου κανονισμού αλλά είδαμε και τι δεν λειτουργεί. Δεν ε, απευθύνομαι σε εσά, γνωρίζω ότι αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης αλλά επιτρέψτε μου να εκφράσω μια τεράστια έκπληξη πάνω σε ένα ζήτημα που δεν προσφέρει στην Ευρώπη τα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα για την καταπολέμηση της κρίσης. Κυρία Χάρκιν, θέλετε να λάβετε το λόγο. Αν μου δώσετε δύο λεπτάκια. Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις και μετά κάποιες απαντήσεις. Ο τελευταίος ομιλητής μιλάει για τη θέση της γερμανικής κυβέρνησης και λέει πως τη νέα μορφή δεν το στηρίζουν. Ανέφερε δύο ζητήματα τη συμπερίληψη των αγροτών και τον ορισμό της κρίσης. Υπάρχουν άλλα ζητήματα που προκαλούν προβλήματα ή αυτά είναι τα βασικά. Αυτό θα ήθελα, αν μπορείτε να μου πείτε. Ναι, ευχαριστώ που κάνετε πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Εγώ είχα καταλάβει πως ήταν ε, η θέση της Γερμανίας ε, ήδη από την αρχή του Ταμείου αλλά τώρα μπορείτε να μας το διευκρινίσετε, κυρία Χούζεμαν. Να πω κάτι για τον ορισμό της κρίσης. Ε, πράγματι τα δύο αυτά σημεία τα ανέφερα είναι σημαντικά, αλλά πιστεύω πως ακόμα και αν ε, κάνει τις διορθώσεις στο Κοινοβούλιο για τη γεωργία, για ένα πιο συγκεκριμένο ορισμό της κρίσης, από όσο ξέρω η γερμανική θέση στο Συμβούλιο δεν θα αλλάξει. Και έχει δίκιο ε, η κυρία Πρόεδρος. Ε, η θέση η γερμανική είναι να σαφές όχι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την παγκοσμιοποίηση. Αυτά. Μα μας επιβεβαιώνεται τον θετικότατο χαρακτήρα της γερμανικής εμπειρίας ε, όταν χρησιμοποίησε τις δυνατότητες κινητοποίησης ε, του συγκεκριμένου ταμείου. Είναι, είναι αστεία η κατάσταση για εμένα ως υπεύθυνο για το Ταμείο. Σας είπα ποια ήταν τα αποτελέσματα που είχαμε. Ε, ξεκαθάρισα επίσης πως αν δείτε ολόκληρο τον τομέα της πολιτικής ε, ε, στον τομέα της εργασίας είπα πως είναι το κερασάκι στην τουρτα και παρουσίασα πως αν δεν το είχαμε θα είχαμε εθνικά μέτρα ε, που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Οπότε αυτά επιβεβαιώνονται και από τις κυβερνήσεις των κρατηδίων αλλά όπως σας είπα υπάρχει αυτή η απόφαση να μην ε, Ευχαριστούμε για τις διευκρινήσεις, ε, ήταν πολύ σημαντικές. Προτού να σταλεί η έκθεση κυρίας Άρκιν στη μετάφραση, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με την Επιτροπή Γεωργίας, πώς θα οργανώσουμε τις εργασίες μου κλπ. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι που μας διαφωτίσατε. Ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσα και ανοιχτή συζήτηση. Το μήνυμα ήταν σαφές ε, σε ό,τι αφορά το γεωργικό θέμα. Τώρα, περνάμε στο σημείο 14. Ο κύριο ε, Νταρντέν έχει το λόγο για την παρουσίαση των τροπολογιών στην γνωμοδότησή του αναφορικά με το πρώτο τμήμα του ΤΟΥΠΑΚ που αφορά την ενίσχυση οικονομική και δημοσιονομική εποπτείας των κρατών μελών τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρέ δυσκολίες αναφορικά με την χρηματοοικονομική του σταθερότητα στη ζώνη ευρώ. Κύριε Νταρντέν, ευχαριστώ Πρόεδρε να περιμένω μερικά δευτερόλεπτα για να επικρατήσει ησυχία. Merci. Euh, Ευχαριστώ. Να πω ότι πολλές τροπολογίες κατατέθηκαν, πάνω κάτω 90 των αριθμών. Ε, έχω καταθέσει και εγώ κάποιες τροπολογίες. Ε, συνολικά οι τροπολογίες αυτές ε, κατά κάποιο τρόπο συμπίπτουν με τις θέσεις μας. Ίσως θα πρέπει να συντάξουμε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες και θα προτείνω στους σκιώδεις ηγητές να συναντηθούμε για να το εξετάσουμε από εκείνο το θέμα αυτών των συμβασικών τροπολογιών. Τώρα, υπάρχει το ζήτημα της αρμοδιότητας, αρμοδιότητας της ε, Επιτροπής μας πάνω σε ορισμένες τροπολογίες ε, που αφορούν ιδιαίτερα την Οικονομική και Νοσβεντική Επιτροπή, ειδικά όταν ε, Μιλάμε για νέες διαδικασίες ε, που θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή ή για κάποιες πλειοψηφίες ε, στο Συμβούλιο. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε τα πράγματα. ώστε η Επιτροπή μας ε, να γνωρίζουμε κατά πόσον μπορεί και πρέπει να αποφανθεί επί των συγκεκριμένων τροπολογιών, εάν θα τις διατηρήσουμε ή εάν θεωρούμε ότι θα πρέπει να τις απορρίψουμε. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Κάτι ακόμα. Είναι ένα ζήτημα που επανέρχεται το θέμα της ε, των μακροοικονομικών προϋποθέσεων ορισμένοι ζητούν την ε, διαγραφή του άρθρου 6 παράγραφος α θα καταθέσει μια τροπολογία που έλεγε ότι αντί να στηριχθούμε στις, ε, πάνω σε ένα κράτος που παρήμενε τις δυσκολίες, θα πρέπει να φροντίσουμε να το βοηθήσουμε αυτό το και όχι να το σπρώξουμε και το βυθίσουμε. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η καλύτερη στρατηγική και κρίνω ότι αυτό θα δημιουργήσει πολλές συζητήσεις. Και κάτι ακόμα, για να τελειώσω, είναι η κατηγορηματική στάση και θέση ε, μελών που καταθέτουν τροπολογία που ζητάει την διαγραφή του κειμένου αυτού του, του ΠΑΚ. Φυσικά εδώ ερχόμαστε στην προσέγγιση που έχουμε να κάνουμε για το 6-pack, το 2-pack και είχα εκφραστεί την ε, προηγούμενη φορά επί του θέματος ε, αυτή τη φορά έχουμε την ευκαιρία να καταρτήσουμε γνωμοδότηση, να δώσουμε στο έγγραφο μια χρειά πιο έντονη σε ό,τι αφορά την ε, τήρηση της στρατηγικής 2020, ειδικά σε θέματα ανάπτυξης κοινωνικών στόχων, απασχόλησης κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να δράξουμε την ευκαιρία και να τονίσουμε αυτά τα σημεία στην γνωμοδότηση. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω κάποιες τροπολογίες που έχω κάνει στην πρόταση Δερντεν. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με αυτά τα οποία προτείνει εδώ πέρα η Επιτροπή. Το πακέτο μπορεί να είναι χρήσιμο γιατί υπάρχουν και χώρες που έχουν ε, προβλήματα πρέπει να παρακολουθηθούν για να κάνουν διαρθρωτικές αλλαγές αλλά και βεβαίως τις απαραίτητες επενδύσεις από τους προϋπολογισμούς τους. Επιπλέον, πράγματι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στην απασχόληση και την ανάπτυξη, αλλά με τρόπο έξυπνο όχι μόνο να γράψουμε σε ένα κομμάτι χαρτί τις λέξεις ανάπτυξη και δουλειές, αλλά να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα στον πραγματικό κόσμο. Συμφωνώ με την παραπομπή δε στο άρθρο 28 της Συνθήκης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Βεβαίως, πέρα από το θεμελιώδες δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων, υπάρχει και το δικαίωμα στην εργασία. Έχω καταθέσει μια τροπολογία και οπωσδήποτε ο εισηγητής που γνωρίζει την σχετική συζήτηση ελπίζω να το λάβει υπόψη. Επίσης είμαι πεπισμένος πως εάν θέλουμε περισσότερη ανάπτυξη και δουλειές πρέπει να έχουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της ευρωπαϊκής ε, διακυβέρνησης. και νομίζω πως αυτή εδώ πέρα η Επιτροπή πρέπει να δώσει το βήμα για το τι πρέπει να γίνει για την οικονομική διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό έχω προσθέσει δύο τροπολογίες. Μία για το ότι διαπιστώνεται πως κάποια κράτη-μέλη ε, έχουν κάποιες συγκεκριμένες απόψεις, οπότε θα έπρεπε να έχουμε μια αντίστροφη ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο για να ευθυγραμμιστεί και το κείμενο. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει διάλογος και με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπάρχει διαφάνεια στην όλη διαδικασία και μια δημοκρατική νομιμοποίηση. Αναμένω λοιπόν τη συνεργασία με τον εισηγητή και με τους υπόλοιπους και ηγητές για να καταλήξουμε σε συμφασμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που θίξατε και που εμπίπτουν ε, σε θέματα που ενδεχόμενα θέλετε να καταθέσετε τροπολογίες στην Επιτροπή Οικονομικών και όχι εδώ. Αυτό που προτείνω λοιπόν είναι η γραμματεία να σας ενημερώσει σχετικά με τις τροπολογίες που δημιουργούν πρόβλημα αρμοδιοτήτων έτσι ώστε να μπορέσετε να κρίνετε κατά πόσον θα τις αποσύρετε και να υποφελθείτε από την προθεσμία κατά των τροπολογιών για να τις καταθέσετε στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Κύριε Τζούμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ήθελα να αναφέρω τώρα τις δικές μας τροπολογίες, ε, καταθέσει τροπολογίες για να εκφράσω το ότι πρέπει να απορρίψουμε την πρόταση της Κομισιόν. Ε, Η άποψή μου είναι πως τα μέτρα αυτά τα οικονομικά και επιτήρησης του προϋπολογισμού μπορούν να φέρουν ακόμα περισσότερα μέτρα λιτότητας. Σκληρά. Αυτά τα πράγματα επηρεάζουν τη καθημερινή ζωή του κόσμου. Οπότε προφανώς πρέπει να λάβουμε υπόψη την σημερινή πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς εφαρμόζονται τα μέτρα λιτότητας και τι σημαίνουν. Αυξάνουν το χρόνο εργασίας, το καθιστούν, ευκολο, καθιστούν ευκολότερες τις απολύσεις και αυτές οι λύσεις θα δημιουργήσουν ανεργία. Ε, άμεσο είναι αυτό το αποτέλεσμα. Δεν θα ε, κάνουν τα πράγματα καλύτερα θα προκαλέσουν μεγαλύτερη ενέργεια και θα κάνουν δυσκολότερη την, την πρόσληψη. Δεδομένης λοιπόν της ε, ύφεσης της οικονομικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα μέτρα αυτά πραγματικά σταματούν οποιαδήποτε πιθανότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας. Ξέρω πως πρέπει να συμβιβάσουμε κάποια πράγματα αλλά ε, είναι πασιφανές. Χωρίς κάποια δράση δεν θα υπάρξει ανάπτυξη. Οπότε, αυτή είναι, αυτή είναι η θέση μας. Απορρίπτουμε τις προτάσεις αυτές. Κυρία Τύρινα. Α, γρήγορα έφτασε η σειρά μου. Κάποια σχόλια για την έκθεση Τάρνταν. Συγγνώμη που δεν παρακολούθησα την παρουσίασή σας αλλά υποθέτω πως οι προτάσεις σας ήταν οι ίδιες για το καθεστώς το ίδιο. Έχουμε τώρα το διπλό πακέτο μετά από το εξαπλό που έρχεται. Και ακολουθούμε την πορεία που έχει καθοριστεί και κατά βάση αφορά τους προϋπολογισμούς, έλεγχο του ελίματος, του χρέους και σχετική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Ναι, δεν φτάνει αυτό, δεν θα λύσει την κρίση, πράγματι, τα λέμε αυτά. Και έχει και στοιχεία ακόμα που είναι ενισχύουν τον οικονομικό κύκλο, θα κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Τούτου λεχθέντος πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ε, ως πολιτικές ομάδες πως θα έρθουν αυτά τα πράγματα, τα θέμε δεν τα θέμε. Το Συμβούλιο μας ζήτησε μάλιστα να επιταχύνουμε την ε, υιοθέτηση. Θα γίνει λοιπόν αυτό. Αυτό το οποίο θεωρώ λοιπόν είναι πως πρέπει να επηρεάσουμε το περιεχόμενο να είναι πιο ισορροπημένο. Και όταν το λέμε εμεί οι πράσινοι, experiencing severe difficulties, which is, ε, which is the report, must also take in... Οπότε πρέπει να λάβει υπόψη πράγματι την ανάπτυξη και τις δουλειές. Δηλαδή και δεν γίνεται μόνο να ασχολούμαστε με τους προπολογισμούς και να μην έχουμε υπόψη και την κοινωνική πτυχή και τους στόχους του 2020. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν εξίσου ε, μεγάλη πειθαρχία ως προς αυτό όπως και ε, προς τη μεριά των δημοσιονομικών. Νομίζω πως θα είναι βελτίωση των εκθέσεων αυτών, εάν το καταφέρουμε ως Επιτροπή, ελπίζω και στην Επιτροπή Οικονομικών. Αυτή είναι η προσέγγισή μας. Ναι, είναι μονόπλευρη ότι συνεχίζουμε αυτή την πορεία. Από την άλλη θα γίνει ούτως ή άλλως. Οπότε γιατί να μην να προσπαθήσουμε να έχει το καλύτερο περιεχόμενο. Και θα πω, ειδικά η έκθεση Ντάρντα μπορεί να είναι χρήσιμη στο πλαίσιο του κανονισμού. Γιατί ε, τι συμβαίνει, ο τομέα αυτό τώρα είναι τελείω ε, χωρί ρύθμιση. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα, η σχέση Κομισιών Ελλάδας δεν ρυθμίζεται κάπου, δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει νομική προστασία. Γιατί οι μισθοί συμπιέζονται και η Κομισιόν κάνει συστάσεις για του μισθού. Και εδώ πέρα έχουμε άρα την ευκαιρία να βάλουμε κοινωνικέ ρήτρε για να σεβαστούμε π.χ. τους μισθού. Οπότε μπορείτε να το δείτε και ω μια ευκαιρία να α, ρυθμίσουμε κάπως τους κανόνες για πράγματα που συμβαίνουν ούτω ή άλλω σε αυτές τις χώρες και προ όφελο των χωρών αυτών. Ε, δείτε το και έτσι. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλοι που να έχουν ζητήσει το λόγο ο κύριο Νταρντέν. Αλλά προηγουμένως, ε, μόνο ότι υπάρχουν πολλά θέματα που αφορούν στην Οικονομική, κοινωνική, ε, την ε, οικονομική και Επιτροπή, να πω οποιαδήποτε και αν είναι η σύγχυση που μπορεί να προκαλείται σε θέματα αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιτροπών ε, κατακλείδει η στρατηγική του εισηγητή στην Οικονομική και Νοσοντική Επιτροπή θα είναι να συμπεριλάβει στην ε, παράγωγη νομοθεσία το περιεχόμενο μιας ε, συνθήκης και το, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι η τύχη αγνοείται διότι την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε πως στην Ιρλανδία η συγκεκριμένη συνθήκη θα τεθεί σε δημοψήφισμα και καταλαβαίνετε ότι η τύχη της ε, συνθήκης ε, δεν είναι διόλου σίγουρη. Έχετε το λόγο, κύριε Νταρντέν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, που διευκρίνησαν το εύρος των τροπολογιών των αλλά και τη σκέψη τους και θα αναφερθώ στην τελευταία παρέμβαση της συνάδελφου Τούρινεν. Θεωρώ ότι θα πρέπει να πούμε ότι επιθυμούμε ένα κείμενο πιο ισόρροπο, γι' αυτό είναι και το νόημα της εκθεσεώς μου να λάβουμε υπόψη ότι, μάλλον να πούμε ότι αυτοί οι στόχοι λαμβάνουν υπόψη τους στόχους 2020, τους κοινωνικούς στόχους, κοινωνικούς ανάπτυξης και αυτούς που αφορούν στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και οι τροπολογίε νομίζω ότι ενδυναμώνουν αυτό το πνεύμα. Θεωρώ πως μπορούμε από αυτού να συμφωνήσουμε. Εάν δεν το πούμε εμείς, και δεν τον βάλουμε στην γνωμοδότησή μας, δεν νομίζω να συμβεί σε καμία άλλη επιτροπή. Γι' αυτό θεωρώ πως πρέπει να ε, μείνουμε σε αυτά τα ζητήματα. Οι συζητήσεις που θα έχουμε με τους ε, σιώδες ηγητές ε, θα με απασχολήσουν. Ευχαριστώ. Καλή εργασία λοιπόν για την σύνταξη των συμβαστικών τροπολογιών. Ξέρω πως η ΕΚΟΝ ε, έχει μεταθέσει το χρονοδιάγραμμά τη, διότι η προθυμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 12η Μαρτίου και η ψηφοφορία θα διεξαχθούν στις 26 Απριλίου. Ναι, γύρω στις 26 Απριλίου δεν είμαι σίγουρη, αλλά κάπου εκεί. Αυτό δεν αλλάζει και πολλά πράγματα στο δικό μας χρονοδιάγραμμα. Θα εξετάσουμε λοιπόν τις συμβασικές τροπολογίες της 29 Φεβρουαρίου. Συγγνώμη, λάθος, λάθος. Θα ψηφίσουμε στις 26. Μάλλον θα τις εξετάσουμε στις 26 θα ψηφίσουμε στις 27. Περνάμε στο σημείο 15 της ημερησίας διατάξεως. Δίνω το λόγο για την έκθεση της κυρίας Φερέρα για τα αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και για τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματο των κρατών μελών ζώνη ευρώ στον εισηγητή μα, κύριο Ντόιτς. Σα ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εξάτιμοι συνάδελφοι. Όπως πριν από μερικές εβδομάδες είχαμε ήδη εξετάσει αυτό το θέμα. Στα πλαίσια του σχεδίου της ε, Κομισιόν του τουλάχιστον. Είπανε ότι εντάξει, είχαμε το 6 pack και τώρα έχουμε το 2 pack. Πρώτα 6, μια δέσμη 6 μέτρα, τώρα 2 μέτρων. Πρόκειται για δύο θέματα που είναι στενά συνδεδεμένα <clears throat> και από τα εξετάζουμε αυτή τη στιγμή από κοινού. Έχουν παρόμοιους στόχους. Πήραμε 80 τροπολογίες για την πρόταση αυτή γνωμοδότησης. Όλες αυτές οι τροπολογίες για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα ήθελα να ευχαριστήσω γιατί όλοι θέλουν να επιτύχουν κάτι καλύτερο. Δεν μπορώ παρά να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι οι περισσότεροι των τροπολογιών αυτών είναι επικοδομητικές και συμφωνούν με τις δικές μου απόψεις. Γι' αυτό μπορούμε να τις υποστηρίξουμε δηλαδή. Μια που βελτιώνουν και συμπληρώνουν το κείμενο. όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τους στόχους ε, στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες τροπολογίες που δεν μπορώ να δεχτώ, είναι σαφές αυτό. διότι θα καθιστούσαν το κείμενο πιο δυσνόητο, ασυνεπές, γιατί καλύπτουν κάποιες θέσεις επίσης, οι οποίες ε, άπτονται του ουσιαστικού τμήματος της πρότασης της Κομισιόν. Με τις περισσότερες, όπως είπα, μπορώ να συμφωνήσω. Αυτό που προτείνεται καθιστά το κείμενο πιο δυσνόητο Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω. Μπορώ να υποστηρίξω εκείνες τις τροπολογίες οι οποίες εξακολουθούν να εντάσσονται στο ίδιο σκεπτικό. Ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχει η ισορροπία μεταξύ των στόχων ε, απασχόλησης και των κοινωνικών στόχων και από την άλλη μεριά των δημοσιονομικών στόχων. Και ότι τελικά ε, ο, η ανεξαρτησία των κρατών μελών για το δημοσιονομικό θέμα θα πρέπει να διατηρηθεί. Να υπάρξει δηλαδή αυτή η ισορροπία που είπαμε. Θα προετοιμάσω βέβαια κάποιες συμβαστικές τροπολογίες, τις οποίες θα υποβάλω στους σκιώδεις και ελπίζω ότι θα υπάρχει δυνατότητα η Επιτροπή μας να δεχθεί τελικά ωραία αυτή την γνωμοδότηση. Πρόεδρος. Ο κύριος Ντεμπάκερ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την πρόταση που υπέβαλε. Όπως και κοινώς έτσι και εγώ σε γενικές γραμμές συμφωνώ με την πρόταση και έχω εδώ κατά νου ε, τις ε, τροπολογίες που θα υποβάλει που πιστεύω ότι θα συμπληρώσουν ε, χρήσιμα το κείμενο. Αυτό σχετίζεται βέβαια με την στρατηγική του 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι καλό που τονίζεται επίσης ο συσχετισμός με το Ευρωπαϊκό Εξόμενο, Ανάπτυξη και Σταθερότητα. Η αναφορά στο άρθρο 9 για να προωθήσει ένα υψηλό επίπεδο απασχόληση η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό, βεβαίω με τρόπο βιώσιμο και στο πλαίσιο τη συζήτηση που γίνεται εδώ πέρα, ε, ίσω και λυσμένων προπολογισμών για να έχουμε μια πραγματική τέτοια πολιτική. Θέλω να τονίσω κάποια πράγματα τα οποία βεβαίω μα απασχολούν Βεβαίως συμφωνούμε με την ανάγκη για περισσότερη απασχόληση και κοινωνική προστασία, αλλά βεβαίως το να δημιουργούμε βέβαιες κοινωνικές ε, θέσεις εργασίας με αυτόν τον τρόπο δεν ε, προσφέρει τίποτα. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ε, ανάπτυξη και απασχόληση με αυτόν τον τρόπο. Επίσης θα πρέπει να γίνουν κάποιες συμπληρώσεις στην ε, πρόταση της Κομισιόν που θα πρέπει να αποτελέσει την βάση μας εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα εγώ να συζητήσουμε σε αυτή την Επιτροπή το εάν χρειαζόμαστε πράγματι ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Διάσωσης πέρα από το ε, ευρωομόλογα για να δούμε αν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη σταθερότητα του μακροοικονομικού συστήματος και η δεύτερη πρόταση που έχω κάνει είναι κράτη-μέλη τα οποία έχουν προβλήματα με τα δημοσιοοικονομικά τους, θα πρέπει βέβαια να ειδοποιούν εγκαίρως την Κομισιόν όσον αφορά την συσσόρευση των χρεών αυτών. Έκανα λοιπόν προτάσεις για μια νέα διάταξη, πως θα πρέπει να είναι οι ε, εθνικοί υπερπολογισμοί ισοσχελισμένοι ή και πλεονασματικοί. Επίσης το, το 3% το οποίο αναφέρεται ως ε, όριο ελλείμματος δεν σημαίνει πως πρέπει να είναι ο κανόνας, θα πρέπει να είναι σε θέση να έχουν ισοσκελισμένους ή ακόμα και πλεονασματικούς προϋπολογισμούς στα κράτη. Επίσης, θα πρέπει να μπορούμε να διδασκόμαστε ο ένας από τον άλλον, να ακούμε στον άλλον. Αυτό οπωσδήποτε είναι απολύτως αναγκαίο. Θα πρέπει λοιπόν και εδώ πέρα αναμένω την ε, συνεργασία με τον συγητή και τους κοιόδες συγητές ε, για να κάνουμε συγκεκριμένε προτάσεις για το διπλό αυτό πακέτο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τουριν. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ που ε, καλέσατε τους σκιώδες να συνεργαστούν. Εγώ για το συνολικό καθεστώς έχω ένα σύντομο σχόλιο. Οικονομική διακυβέρνηση, ναι, αλλά οπωσδήποτε συσσωροπημένη. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε με αυτές τις δύο εκθέσεις. Δηλαδή όχι μόνο ε, διακυβέρνηση που βασίζεται στο ελλείμματα και στα χρέη, αλλά στις επενδύσεις, ε, στις ε, δεσμεύσεις για την Ευρώπη 2020 και πιο εξισορροπημένη διακυβέρνηση από ό,τι που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μας, τον, τους πράσινους, που έχουμε τονίσει και θα που το συνεχίζουμε να τονίζουμε, είναι το θέμα του δημοκρατικού ελέγχου. Γιατί άμα δίνονται αρμοδιότητες και εξουσίες στο ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει σωστός Δημοκρατικός έλεγχος είναι η δυνατότητα του σώματος εδώ να παρέμβει, των κοινωνικών εταίρων και των ε, σημαντικών ε, μη κυβερνικών οργανώσεων. Αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Κάτι άλλο, και το έχουμε κάπως προσθέσει εδώ, θα πρέπει να υπάρχει και μία αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων. Όταν δηλαδή υπάρχουν κάποιες συστάσεις ε, προς τα κράτη-μέλη, θα πρέπει και θα είναι υποχρέωση της Κομισιόν να εξεταστούν οι κοινωνικέ επιπτώσει. Δεν το έχουμε αναπτύξει το θέμα, αλλά θα μπορούσαμε ίσως να αναπτύξουμε τι σημαίνει η αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων. Ανεργία, φερρυπίν, ε, κοινωνικά ωφέλη και κοινωνικά επιδόματα, ε, κοινωνικός αποκλεισμός, φτώχεια και μισθή. Θα πρέπει λοιπόν να περιλάβουμε τι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την κοινωνική ε, αξιολόγηση που είναι πάρα πολύ σημαντική όπως και το θέμα του δημοκρατικού ελέγχου και της εξορρόψης. Προσβλέπουμε λοιπόν στην περαιτέρω συνεργασία. Και θα επαναλάβω αυτό που είπε ο κ. Ζαρτάν, ότι η Επιτροπή ε, μας εδώ έχει όχι μόνο ε, δικαίωμα, αλλά υποχρέωση να τονίσει ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή το θέμα ότι οι οικονομικές πολιτικές της Ένωσης θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Αλλιώς τι κάνουμε εδώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο λόγια. Να σας πω ότι η οι τροπολογίες που υποβάλαμε για την έκθεση αυτή είχαν σαν στόχο την συνοχή μεταξύ των δύο κειμένων. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό να υπάρχει συνοχή μεταξύ των δύο αυτών κειμένων μέσα στο ίδιο σκεπτικό που περιγράφει αυτή τη στιγμή να υπάρχουν δηλαδή εξορροπημένες δημοσιονομικές ε, πολιτικές ε, που θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη είτε βράχη είτε μακροπρόθεσμα την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τον κύριο στόχο της ε, καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Έχουμε υποβάλει σχετικές τροπολογίες και βέβαια είμαστε σε συνδυάσεις του συγγητή να τις συζητήσουμε μαζί του. Ευχαριστώ, ο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Πρέπει να ε, παραδεχτώ κάτι, είμαι μεγάλος οπαδός του Τούπακ. Για να αποφύγουμε εδώ πέρα τις παρεξηγήσεις, δεν εννοώ βεβαίω τις προτάσεις αυτές, αλλά ξέρετε το, το γνωστό ράπερε τον Τούπακ Σακούρ που σκοτώθηκε πριν από χρόνια. Οπότε όταν λέω Οπότε δεν θέλω, εν πάση περιπτώσει, και το δικό μας το Τούπακ εδώ πέρα να συναντήσει τη, το ίδιο, να έχει το ίδιο τέλος του Τούπακ σε ως χωρέστονα. Πρέπει λοιπόν να επιτευχθεί μια ισορροπία για να μην σκοτωθούν και πεθάνουν άδοξα αυτές οι προτάσεις πρέπει να μειωθούν πράγματι τα ελλείμματα των προϋπολογισμών αλλά να υπάρχει και μια ισορροπία των στόχων όσον αφορά την ε, απασχόληση και τα κοινωνικά. Οπότε χαιρετίζω τις τροπολογίες των συναδέλφων και θα προσπαθήσω να δημιουργήσω μια ξεκάθαρη γραμμή για να επιτύχουμε μια συνένεση. Θα υπόκειστε λοιπόν στο ίδιο καθεστώς ε, σε αφορά το διάγραμμα με αυτό του κυρίου Dark δηλαδή ότι με βάση τις τρο... τροπολογίε τροπολογίες που θα εξετάσουμε στι 26 Μαρτίου θα ψηφίσουμε στι 27. Και φτάνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο σημείο της μεσή διατάξεω. Υπάρχουν 140 τροπολογίε ε, αισίω που κατέθεσαν στη γνωμοδότηση τη κυρία Ζήμερ Πρόκειται για μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Γυναικών σχετικά με τις ίσες αμοιβέ για ίση εργασία. Κυρία Συγκήτρια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι αναφέρατε πως έχουν κατατεθεί 140 τροπολογίες. 140 από όλες τις ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό σπάνιο. Υπάρχουν τροπολογίες από βουλευτές που δεν είναι ε, μέλη της Επιτροπής μας. Υπάρχουν και άλλες ε, τροπολογίες από συναδέλφους που είναι μέλη και αυτής της Επιτροπής και της Επιτροπής Γυναικών. Και θεωρώ πως θα πρέπει να έχουμε μία συνέπεια εδώ πέρα στους στόχους για τη γνωμοδότησή μας αλλά και για τη σύνταξη βεβαίως της ε, έκθεσης αυτής. Είχα αυτή την εβδομάδα την, επιτρο... την δυνατότητα να είμαι παρούσα στη συζήτηση στην Επιτροπή Γυναικών και ε, έλαβα υπόψη την τοποθέτησή τους και μπορώ να πω πως εξετάζοντας τροπολογίες αυτές θα νομίζω μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε μεγάλο βαθμό για τις τροπολογίες τώρα. Εγώ ίδια κατέθεσα 14 από αυτές. Αυτό βεβαίως σχετίζεται κυρίως με το ότι η γνωμοδότηση ε, βεβαίως ε, πρέπει να είναι αρκετά σύντομη, γι' αυτό είχα, είχα στόχο να την κάνω μετά ε, πιο λεπτομερή. Νομίζω πως έχουμε ούτως ή άλλως τους ίδιους στόχους, ε, αυτό είναι καλό. Είναι νομίζω ζήτημα απλά εφαρμογής εδώ πέρα αυτό το οποίο μας απασχολεί. Ε, δηλαδή να πάνε στις, στα ανάλογα άρθρα ή ανάλογες τροπολογίες πάνε εκεί που αντιστοιχούν. Και να δούμε βέβαια πώς μπορούμε να τα συνοψίσουμε όλα αυτά σε κάποιες συμβιβαστικές ε, τροπολογίες. Θα προσκαλέσω τους ή άλλους τους κοιόδους την ερχόμενη εβδομάδα σε μία συζήτηση, να δούμε δηλαδή πώς θα συμβαστεί καλύτερα η επαγγελματική ζωή, η μερική εργασία η ε, επισφαλής εργασία, να μην υπάρχει εκεί πέρα ε, πρόβλημα στις συντάξεις μετά. Βεβαίω να μην υπάρχει ανισότητα με βάση το φύλλο. Αυτό το λέω γιατί υπήρξαν νέα στατιστικά στοιχεία από τη Eurostat που οδηγεί στο ότι ε, πρέπει να γίνει μια διόρθωση στο σχέδιό μας, γιατί είχαμε τα νούμερα του 2009, τώρα έχουμε τα νούμερα του 2010, οπότε γίνεται λόγος για ένα 16,4% συνολικά όμως μιλάμε για 16,8% στις χώρες του ευρώ Κατά την άποψή μου αυτό οφείλεται στο ότι παραδείγματο χάρη η Πολωνία είναι τώρα στο 1,9% δηλαδή είχαμε μια σημαντική μείωση ε, του μισθολογικού χάσματος ε, οπότε είναι ακριβώς το ζήτημα των κριτηρίων και των στατιστικών στοιχείων που χρησιμοποιούμε. Οπότε θα πρέπει να έχουμε πραγματικά συγκρίσιμα ε, στοιχεία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι θα ήθελα ακόμα να πω. Η κυρία Στάινρουκ πρότεινε η, η Ευρωπαϊκή ημέρα ίσης πληρωμής που προβλέπεται για αύριο να συνδεθεί με μία ημέρα δράσης. Εδώ πέρα παραπέμπω στο πρόβλημα πως σε όλα τα κράτη-μέλη υπάρχουν τελείως διαφορετικά δεδομένα, δηλαδή de facto δεν υπάρχει ε, μία ευρωπαϊκή ημέρα ίσης αμοιβή για ίδια δουλειά Οπότε μπορούμε να κάνουμε, καταθέσουμε μια προφορική τροπολογία και να απαιτήσουμε, αν θέμε να είμαστε αποτελεσματικοί, ε, τουλάχιστον να γίνεται εκδήλωση την ίδια μέρα. Υπάρχουν και τροπολογίες που αναφέρονται στην ε, λεγόμενη ευέλιξη ασφάλεια περισσότεροι δεν αμφισβητούν αυτή την έννοια σε αντίθεση με εμένα. Να, ούτως ή άλλως θα γίνουν οι ψηφοφορίες οι σχετικές από κάποιους βουλευτές ε, από έναν βουλευτή υπάρχουν τροπολογίες που είναι αντίθετες με όλων των υπολείπων ε, είμαι σίγουροι πως δεν θα υπερψηφιστούν θα, θα τα δούμε αυτά στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ε, Η κυρία Εστρέλα και θα ακολουθεί ο κύριος Κουστόφσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόμαλος της Σοσιαλιστικής Ομάδας θα ήθελα να πω πως ε, στην ουσία συμφωνούμε με τις ε, προτάσεις που έχουν υποβάλει οι συνάδελφοι. Υπάρχουν όμως και κάποιες προτάσεις με τις οποίες διαφωνούμε. Χρειάζεται να εργαστούμε και εμείς είμαστε διαδεθειμένοι να συνεργαστούμε με την εισηγήτρια ώστε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές λύσεις, κάτι που θα καταστήσει και πιο απλές τι ψηφοφορίε και θα προσφέρουν μεγαλύτερη συνοχή και συνέπεια στο κείμενο το οποίο θα αποσταλεί στην αρμόδια επί Επιτροπή, Επιτροπή Γυναικών. Το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Η εισηγήτρια δήλωσε πως ε, έχει επιτευχθεί αφενός πρόοδος και αφετέρου οπισθοδρόμηση μέχρι 2009-2010 ε, ε, σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurostat είδαμε ότι περάσαμε από το 17,5% σε 16,4% ε, δεν είναι και τεράστια η διαφορά αλλά το 2005 αυτή η διαφορά ήταν μικρότερη, ήταν της τάξης του 15% σε της αφορά αμοιβές ανδρών γυναικών. Ε, αυτό είναι σημαντικό, είναι σοβαρό. Είναι ένας αγώνας που πρέπει να συνεχίσουμε διότι διαπιστώνουμε ότι δεν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος και μία πάμε μπρο, μία πάμε πίσω. Έχουμε καταθέσει κάποιες τροπολογίες για να προαγάγουμε τις βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έτσι ώστε και οι επιχειρήσεις ε, να έχουν κίνητρα για να βελτιώσουν την συμπεριφορά τους. Διαφορετικά θα πρέπει να εφίστανται κυρώσεις ε, όταν εφαρμόζουν απαράδεκτες, ε, απαράδεκτη διακριτική μεταχείριση. Γνωρίζουμε παραδείγματος χάρη πως οι γυναίκες γενικά θίγονται και σε ζητήματα σταδιοδρομίας πλήττονται συχνά. Πολλές φορές δεν ε, λαμβάνουν ε, και ε, πριν αποδοτικότητας. Παραδείγματος χάρη όταν βρίσκονται σε άδεια μητρότητας δεν λαμβάνουν αυτά τα πριν. Κάτι άλλο σχετικά με τα συστήματα αμοιβή. Αυτά τα συστήματα θα έπρεπε να είναι πιο διαφανή και να υπάρχει πρόσβαση από πλευρά κοινού, διότι γνωρίζουμε ότι στον δημόσιο τομέα, εντάξει, είναι εύκολο να γνωρίζουμε το βαθμολόγιο, αλλά και τις αμοιβέ, αλλά στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει έλλειψη διαφάνειας και ούτε οι διεργαζόμενοι στην επιχείρηση δεν γνωρίζουν ποιες ε, είναι οι αμοιβέ ε, των συναδέλφων και αυτό όπως καταλαβαίνετε εμποδίζει το να έχουμε στοιχεία περί αμοιβών. Τώρα η μεθοδολογία συλλογής ε, δεδομένων δεν είναι η αυτή σε όλα τα κράτη-μέλη και έτσι δεν γνωρίζουμε μέχρι ποιο σημείο Κάποιες πρόοδοι είναι πραγματικές και ουσιαστικές. Πάντως ε, πρέπει να καταγράψουμε τα θετικά βήματα τα οποία έχουν γίνει στην Πολωνία, παραδείγματος χάρη, όπου εκεί έγινε όχι ένα βήμα, ένα άλμα θα λέγαμε. Και για να καταλήξω, θεωρώ πως έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε πως ε, η ωριαία αμοιβή δεν είναι το μοναδικό στοιχείο για αξιολόγηση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και κάποια επιδόματα που χορηγούνται σε ορισμένους εργαζόμενους και όχι σε άλλους. Και αυτά τα επιδόματα οδηγούν σε υψηλότερες αμοιβές. Οι γυναίκες είναι η ομάδα που έχει συνήθως επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, ε, εργάζεται με μερική απασχόληση κλπ. Και αυτό συμβάλλει στο να υφίστανται κυρώσεις ε, στον τομέα των αμοιβών ε, οι γυναίκες. Έχουμε λοιπόν δυνατότητα να υποβάλουμε προτάσεις που θα στοχεύουν στην καταπολέμηση της άνησης αμοιβής μεταξύ ανδρών Αυτή είναι μια πολύ παλιά ιστορία που ξεκίνησε αρχάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχή της Ισαμβής είναι μια αρχή η οποία θεσπίστηκε το 57. Ευχαριστώ κ. Ε, ναι, Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Μιλάω βέβαια εξ ονόματος ε, της συναδέλφου της κυρίας Σουμπλεύσκα που είναι σκιώδης συγγήτρια, αλλά δυστυχώς απουσιάζει. Η γνωμοδότηση έχει ως ε, Η συνάδελφος ε, θεωρεί τις τροπολογίες θετικές. Βεβαίως κάποιες επαναλήψεις δεν μπόρεσαν να αποφευχθούν, αλλά ελπίζω πως οι συμβαστικές τροπολογίες κυρία Τσίμερ θα κάνουν το κείμενο πιο συνεκτικό. Εγώ θα προτείνω η πολιτική μου ομάδα να στηρίξει τις ε, περισσότερες ε, τροπολογίες. Ε, τώρα όσον αφορά τις κυρώσεις που προβλέπονται για τους επιχειρηματίες. Αυτές προβλέπονται ούτω ή άλλω από τον νόμο. Μπορεί να πάει κάποιο στα δικαστήρια. Αυτό το οποίο στηρίζουμε εμείς είναι διοικητικέ κυρώσεις που μπορούμε να προτείνουμε. Επίσης στηρίζουμε την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά την ιδέα της ε, ίσης ε, πληρωμής, αλλά δεν είμαι σίγουρος πως πρέπει να κατακαιρματιστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοτεχνικό Ταμείο και να ασχολείται με ζητήματα αμοιβών. Προτείνω η ομάδα μου να συζητήσει τις νέες νομοθετικές προτάσεις που θα προτείνει η Κομισιόν. Κύριε Ήρσφη. Ευχαριστώ. Κάθε χρόνο έχουμε το θέμα αυτό, γιατί δεν έχει λυθεί. Είναι θλιβερό αυτό. παρόλα όλα αυτά, είναι θέμα με πολλές πτυχές. Και βεβαίως οφείλεται στο ότι οι γυναίκες έχουν τα επαγγέλματα εκείνα τα οποία εκ των προτέρων πληρώνονται λιγότερα και πρέπει να δούμε και την πτυχή της φτώχειας που συνεχίζεται και στη σύνταξη. Τώρα συγκεκριμένα για το θέμα μας εδώ πέρα. Οπωσδήποτε σημαντική πτυχή είναι πως πολλές γυναίκες εργάζονται σε χαμηλόμιστες δουλειές, αλλά και σε γυναίκες με προσόντα βλέπουμε αυτή την απόσταση. Και, άρα, ισχύει και εδώ πέρα, ε, θα πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα κινήτρων. Οι επιχειρήσεις θα εξαρτηθούν περισσότερο από τις γυναίκες για δημογραφικούς λόγους. Οπότε θα πρέπει και οι γυναίκες να μπορούν να ε, το διαφημίσουν, ότι πληρώνουν την ίδιο μισθό. Για να μπορούν να πάνε και οι γυναίκες σε αυτές τις επιχειρήσεις. Έτσι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα κινήτρων να πούμε ναι, θέλουμε γυναίκες με ε, προσόντα και μας ενδιαφέρει να πληρώνονται ε, με τον ίδιο μισθό. Και δεν ανάγκη πάντα να υπάρχουν, ε, να είναι κυρώσεις αυτά τα κίνητρα. Η κυρία Μχάρκιν και μετά η κυρία Κορνέλισεν. Ευχαριστώ. θα σας διαβάσω και εγώ την άποψη μια συναδέλφου. Είπε να ευχαριστήσω λοιπόν την κυρία Τσίμερ και να κάνω δύο γενικά σχόλια. Είναι μεγάλο το χάσμα πράγματι, αλλά με βάση τα σατσικά στοιχεία που έχουμε σήμερα, μπορούμε να συγκρίνουμε το μόνο το ωριαίο εισόδημα. Αλλά ο στόχος μας είναι να έχουμε ίδιες πηγές, ίδια πληρωμή για ίδια δουλειά για να κλείσει το χάος. Οπότε σας προσκαλώ λοιπόν εδώ πέρα να απαιτήσουμε στατιστικά στοιχεία που περιγράφει το χάσμα ή την πληρωμή ανδρών και γυναικών για την ίδια δουλειά, ίδιας αξίας. Θα πρέπει να παρακολουθούν αυτά τα στοιχεία τα κράτη-μέλη και όχι γενικώ το ωριαίο εισόδημα. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω, αν ε, ερχόμαστε έτσι κοντά στον στόχο μας, ε, ο οποίος είναι αυτός τον οποίο περιέγραψα. Και πάλι ευχαριστούμε την κυρία Τσίμερ. Κυρία Κορνέλισεν. <clears throat> Yeah, uh, is... Η έκθεση αυτή ε, αποτελεί εν μέρει μια επανάληψη έκθεση που είχε γίνει την τελευταία θητεία του Κοινοβουλίου. Η Κομισιόν όμως δεν αντέδρασε τότε και τότε είχαμε ζητήσει κατευθύνες γραμμές ε, και μεγαλύτερη δράση σε νομοθετικό επίπεδο. Αλλά εντωμεταξύ έφτασε η συνδίκη της Λισαβόνας ε, που μας δίνει κάποια δικαίωμα πρωτοβουλία το οποίο και θα χρησιμοποιήσουμε μέσω αυτού, αυτής της έκθεσης. Για το περιεχόμενο όλοι συμφωνούμε ότι η διαφορά αμοιβών ε, ε, μας απασχολεί. Βλέπουμε ότι δεν συγκλίνει. Άρα χρειάζονται περισσότερη δράση να αναλυφθεί. Έχουμε καταθέσει μόνο μία τροπολογία όπου ζητάμε από την Κομισιόν στεναρά να αντιδράσει αυτή τη φορά. Ελπίζουμε πως η τροπολογία αυτή θα υποστηριχθεί. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να στηρίξουμε και τις τροπολογίες σας. Η εισηγήτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Να αναφερθώ σε εσάς κύριε Κορνέλησεν Ναι, βεβαίως. Θα στηρίξω όλες τις τροπολογίες που βασίζουν σε... Ε, απαιτούν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα που θα ξεκαθαρίζουν πως τελείωσε η υπομονή μας με την Κομισιόν. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Ε, άκουσα την Κομισιόν στην Επιτροπή Γυναικών που αναφέρθηκε στην έκθεση της κυρίας Μπάουερ. Και πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Η έκθεση είναι έτσι δομημένη ώστε μας δίνει τη δυνατότητα να προβούμε σε περαιτέρω διευκρινήσεις ε, εάν αυτό απαιτείται εκ των προτέρων έχει σχεδιαστεί έτσι και πολλές ιδέες και πρωτοβουλίες με βρίσκουν σύμφωνοι π.χ. αυτή της κυρίας Χίρς είναι πολύ ενδιαφέρουσα να πούμε δηλαδή ότι δεν θέμε μόνο κυρώσεις που εγώ πιστεύω ότι χρειάζονται αλλά και ένα θετικό στοιχείο και να πούμε οι επιχειρήσεις που είναι δραστήριες και υπεύθυνε γιατί να μην τις διαφημίσουμε κιόλας. Να δώσουμε ένα βραβείο. Um, kleines bisschen etwas jetzt äh, ganz am Anfang. Δεν ξέρω, υπήρχε μια παρεξήγηση με αυτά τα οποία είπε η κυρία Κοίταξα τις ε, ε, τροπολογίες σας. Δεν είναι μία τροπολογία για να συμβιβαστούμε. Πρέπει να δούμε και τις υπόλοιπες τροπολογίες. Να βρούμε δηλαδή συμβασμούς για να έχουμε μία κοινή διατύπωση. Εδώ πέρα συμφωνούμε. για να πετύχουμε μια έκθεση που θα είναι θέση της Επιτροπής. Κύριε Χάρκιν, το ερώτημά σας. Πρέπει να πάμε και πιο κοντά στη, λύση του προβλήματος. Αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε και θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, οπωσδήποτε προσεχώς. Αλλά είναι και ευθύνη μας κοινοβουλευτική και γυναικεία, εάν θέλετε, να πούμε ξεκάθαρα πως έχουμε την άποψή μας και δεν θα αφήσουμε την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να κάνουν ό,τι θέλουν. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Την ερχόμενη εβδομάδα θα αποστείλω πρόσκληση για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. 26 Μαρτίου θα συζητήσουμε και 27 θα ψηφίσουμε. Και έτσι η Επιτροπή Γυναικών θα αποκτήσει επιτέλους τη γνωμοδότησή μας για την Ολομέλεια του Μαΐου 2. Ολοκληρώσαμε 26-27 Μαρτίου το Επανειδήν.